So, I would like, please. oh, it's amazing. This is your first leadership it's, it's crazy. So, please, I'm going to. Παρακαλώ, θα ξεκινήσουμε. Ναι, λίγο ησυχία. A bit discipline. so. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση. Καλώς ορίσατε κύριε Τίμερμαντς. Είναι συνεδρία της Επιτροπής ΕΜΒΗ με συνδεδεμένη Επιτροπή την Ήτρε, την, καθώς επίσης και την Άγκρη και Κουλ, τόσο προσκεκλημένες επιτροπές. Θα συνεχίσω γαλλικά. Γνωρίζετε τους κανόνες του παιχνιδιού. 25 ερωτήσεις, 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ερώτηση και 45 δευτερόλεπτα για συμπληρωματική ερώτηση, ε, αν θεωρείτε ότι χρειάζεται. Ε, αυτό βέβαια μετά από 15 λεπτά εισαγωγικής παρουσίασης του κυρίου Τίμερμανς. Δύο λόγια τώρα για να υπενθυμίσω λίγο το χαρτοφυλάκιο του πρώτου εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι αρμόδιος για το κλίμα βεβαίως, αλλά ε, στο χαρτοφυλάκιο του Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας, έχουμε τις μεταφορές, το περιβάλλον, τους ωκεανούς, την ενέργεια, την υγεία, τη γεωργία και τη συνοχή, που σημαίνει ότι, κύριε Τίμερμαν, ουσιαστικά έχετε ε, υπό το Green Deal τα δύο τρίτα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν ε, πολλοί στην Επιτροπή ΕΜΒΗ που χαιρετήσαμε αυτή την αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και διαπιστώσαμε και στις γραπτές ε, απαντήσεις που δώσατε στις γραπτές μας ερωτήσεις κάποια σημεία επί των οποίων θα ήθελα να επιμείνω ιδιαιτέρως όσον αφορά τις προθέσεις σας. Δεσμεύεστε να κάνετε κάποιες προσαρμογές οι οποίες είναι στοχευμένες για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο Επικαλείστε βεβαίως ε, την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία για πρώτη φορά είναι υπό τη σκέπη του Green Deal και Ήσασταν και ιδιαίτερα δραστήριο στη Νέα Υόρκη σε θέματα αποψήλωση δασών. Ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντο έχει ήδη αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε επί του ζητήματο και φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε όσον αφορά τι προθέσει σα. Ολοκληρώνω αυτή την εισαγωγή υπενθυμίζοντα ε, τι, τι λέει ο θείος του spider Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτός ο υπερήρωας στο σινεμά. Ε, ο θείος του Spider-Man λοιπόν έλεγε ότι με τη μεγάλη εξουσία ακολουθούν και μεγάλες ευθύνες. Έχετε λοιπόν πολλές εξουσίες και τώρα πρέπει να αναλάβετε πολλές ευθύνες και έχετε το λόγο για ένα τέταρτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σκοπεύω να ολοκληρήσω όμως ε, όπως κατέληξε και ο θείος Μπεν. Ε, το είδαμε στην αρχή της ταινίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την εισαγωγή. Ε, ελάχιστα έχω να προσθέσω, αλλά θα κάνω μια απόπειρα. Αξιότιμα μέλη, πραγματικά ανέμενα με ενδιαφέρον τη σημερινή μας συζήτηση, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και έχω έρθει σήμερα εδώ για να λάβω την υποστήριξή σας αλλά και την καθοδήγησή σας. Όλοι μας λοιπόν εδώ σήμερα ήμασταν ε, υποψήφιοι στις ευρωεκλογέ του Μαΐου. Απευθυνθήκαμε στους πολίτες μας με τα σχέδιά μας για το μέλλον και τώρα εσείς οι άμεσα αρετοί εκπρόσωποι των πολιτών θα έχετε πέντε χρόνια στη διάθεσή σας έτσι ώστε να μετατρέψετε αυτά τα σχέδια σε πραγματικότητα. Και εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ ελπίζοντας ότι θα με υποστηρίξετε έτσι ώστε να κάνω κι εγώ ε, ό,τι μπορώ από τη δική μου πλευρά στο πλαίσιο τη Επιτροπή Φόντερ Λάιν, ούτω ώστε να ανταποκριθούμε στι υποσχέσει μα. Αλλά το να λέω τώρα εγώ ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο είναι βέβαια ε, ε, τίποτα ιδιαίτερο, γιατί πραγματικά είναι υπαρξιακή ε, φύση η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, πρόκειται για μια επανεκκίνηση, αν θέλετε, τη κοινωνία μα, έτσι ώστε ε, να διατηρήσουμε όσα είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για εμά και να ε, βελτιώσουμε το μέλλον και για τα παιδιά και για τα εγγόνια μα και τι μελλοντικέ γενιέ. Δεν μπορούμε λοιπόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα θαλασσώσουμε. Και βέβαια, δεν θα προβώ τώρα σε ιδιαίτερε διαγνώσει ω προ τα όσα συμβαίνουν, γιατί το να επαναλάβω τα επιστημονικά δεδομένα σε εσά είναι σπατάλη του χρόνου για όλου μα, γιατί όλοι μα γνωρίζουμε τα προβλήματα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και όλοι γνωρίζουμε δηλαδή τι πολύ δυσμενεί συνέπειε που μπορούν να υπάρξουν για τα οικοσυστήματά μα, την υγεία μα και το μέλλον μα. Και γνωρίζουμε όλοι μα ότι οι πολίτε μα θέλουν να αναλάβουμε δράση. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, να αναλάβουμε δράση. Δηλαδή, οι πολίτε θέλουν η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να ενεργοποιηθεί σε επίπεδο αντίστοιχο με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Και επίση ε, θέλουν να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε να ε, ανταποκριθούμε στις καθημερινές πρακτικές προκλήσεις, δηλαδή να έχουν τα τρόφιμα που χρειάζονται, να θερμαίνουν τις κατοικίε τους, να έχουν μια θέση εργασίας, να έχουν ένα καλό σχολείο για τα παιδιά τους, καλή φροντίδα για τους γονείς τους και γενικότερα να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Ο κόσμος λοιπόν και ο κόσμος των πολιτών μας είναι το ίδιο και το αυτό. Μπορούμε δηλαδή να επιτύχουμε μόνο αν φροντίσουμε και τα δύο. Αν το ένα από τα δύο δεν το φροντίσουμε, δεν θα πετύχουμε σε κανένα από τα δύο. Και γι' αυτό λοιπόν εμεί, αν αποφασίσετε να επιβεβαιώσετε την Επιτροπή Φόντερ Λάιν, θα διασφαλίσουμε ότι αυτό ο μετασχηματισμό ε, βαθέων που θα πρέπει να λάβει η χώρα θα είναι και μια δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή, αυτό ο δίκαιο χαρακτήρα θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών μα και θα βασίσουμε τι μελλοντικέ μα εργασίε ακριβώ σε αυτέ τι αρχέ τη δίκαιη μετάβαση. Και θα υπάρξει και ένα ταμείο, ένα αποκλειστικό ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε του ανθρώπου και τι περιοχέ και τι κοινότητε που θα πληγούν περισσότερο ειδικότητα τη βιομηχανικέ τη εξόρισης άνθρακα και τι ενεργοβόρε ε, περιοχέ. Και βέβαια αποτελεί δικό μα καθήκον να καταδείξουμε στου ε, πολιτέ μα ότι το Green Deal, η Πράσινη Συμφωνία, μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή. Και τώρα, όχι σε 50 χρόνια. Ε, δηλαδή, η καθαρότερο αέρα και καθαρότερα ύδατα στα ποτάμια και στου ωκεανού μα είναι αυτό που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμο μέλλον για όλη την ε, ανθρωπότητα. Και βέβαια με οικονομία η οποία θα αναπτύσσεται προ όφελο όλων, όχι μόνο μερικών, και με θέσει εργασία για όλου. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να θέσει ε, την Ευρώπη στο σωστό άξονα, στη σωστή άγουσα, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον, διασφαλίζοντα ότι όλοι θα συμμετάσχουν και κανένα δεν θα μείνει απ' έξω. Ε, και η φιλοδοξία μα είναι βέβαια να είμαστε η πρώτη ήπειρο που θα έχει μηδενικέ εκπομπέ και μπορούμε να το επιτύχουμε έω το 2050 αν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό και την ανάλυση δράση από τώρα. Και τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικά. Δηλαδή, εγώ θα προτείνω μια νομοθεσία για το κλίμα μέσα σε 100 μέρε από την ανάληψη τη θητεία μου, έτσι ώστε να υπάρξει κατοχυρωμένη νομοθεσία σε ό,τι αφορά αυτό το φιλόδοξο στόχο του 2050 ε, και να θέσουμε με αυτόν τον τρόπο και την μακροπρόθεσμη, το μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Και από εκεί και μετά θα θέσω υψηλό επίπεδο φιλοδοξία έω το 2030 και θα κάνω νομοθετικέ προτάσει, ώστε να μειωθούν οι εκπομπέ κατά τουλάχιστον 50% ή ακόμα καλύτερα κατά 55%. Επίση, θα επανεξετάσω εξετάσουμε και να θεωρήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια. Και επίση θα πρέπει να ε, είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούμε συμπληρωματικά μέτρα έτσι ώστε να έχουμε καθαρότερε μεταφορέ, λιγότερο ενεργοβόρο ακτήρια και ένα πιο βιώσιμο σύστημα παραγωγή τροφίμων. Δεν έχουμε βέβαια την ε, πολυτέλεια να επαναπαυτούμε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα χρειαστεί να απελπιστούμε, γιατί αν συγκρίνουμε τα πράγματα με το 1990, έχουμε μειώσει κατά 22% τις εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου μα ενώ η οικονομία μα έχει αναπτυχθεί κατά 58%. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί κάτι βλαβερό για την ευρωπαϊκή ε, οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να ανεβάσουμε τώρα τον πύχη, να το θέσουμε πιο ψηλά και να έχουμε ψηλότερη φιλοδοξία. Και έχουμε ε, τις απαραίτητες δεξιότητες, τη γνώση στους ανθρώπους αλλά και την πολιτική βούληση σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τώρα θα μπορούσα βέβαια να αναφέρω και πιο στόχους, ε, ποσοστά, την ε, διεύρυνση του συστήματο εμπορία εκπομπών, αλλά καταρχήν επιτρέψτε μου να σα πω το τι μπορεί να κάνει η Πράσινη Συμφωνία για του πολίτε μα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά του ενίκου των κοινωνικών κατοικιών ε, και του ιδιοκτήτε ε, κατοικιών, ειδικότερα εκείνου οι οποίοι έχουν προβλήματα για να πληρώσουν του λογαριασμού ρεύματό του σήμερα. Αναφέρομαι σε 50 εκατομμύρια Ευρωπαίου σήμερα πολίτε, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αυξηθεί ο λογαριασμό ρεύματό του, θα πρέπει να χαμηλώσει και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Δηλαδή, από κοινού τα κράτη-μέλη με του ε, οργανισμού τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εξεταστούμε ε, ευρύτερα, μεγαλύτερα project ανακαίνιση, έτσι ώστε για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε, να, να έχουμε περισσότερη θερμομόνωση ή με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα συστήματα χρηματοδότηση, έτσι ώστε αυτοί οι πολίτε ε, να ε, να μην χρειάζεται να προκαταβάλουν χιλιάδε ευρώ. Αντιθέτω, θα πρέπει είτε να έχουμε επενδύσει είτε να παράσχουμε επιστοτικέ γραμμέ, έτσι ώστε ε, με ε, του πόρου που θα απελευθερωθούν να καλυφθούν αυτά τα κόστη. Και ε, με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ε, άνετο κατοικίε και χαμηλότερους λογαριασμούς. Όλοι δηλαδή θα υποφεληθούν. Και το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και σε σχέση με σχολεία και νοσοκομεία. Γιατί με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητα θα έχουμε περισσότερα χρήματα ε, και για την ε, παιδεία, για παράδειγμα, και για την ε, δημόσια υγεία, ενώ ε, ταυτόχρονα δημιουργούμε και σταθερές θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν εθνικές πρωτοβουλίες και τοπικές θέσει εργασία. Με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και ευρωπαϊκά υποστηρικτικά προγράμματα με ε, κοινή ε, χρηστογνώσεων και ικανοτήτων μπορούμε να έχουμε μια πράσινη συμφωνία η οποία θα αποβεί προς όφελος των πολιτών. Επίσης, οι πολίτες μας, ε, παρότι για μένα ολοένα και περισσότερο σε πόλεις, διαβιούν την ελεύθερο του χρόνου ε, στη φύση και ανησυχούν για τα όσα συμβαίνουν σε διάφορε γωνιέ του κόσμου. Είτε πρόκειται δηλαδή για τα πτηνάκια στι μέλισσε στην ύπεθρό μα, είτε ε, για τα ψάρια για παράδειγμα και τα ευαίσθητα κοράλια ε, στου ωκεανού, ή τα πλούσια δάση μα και τα άγρια ζώα μα, Όλα αυτά τα εξαφανίζουμε, όλα τα σκοτώνουμε και πραγματικά με ένα πολύ ανησυχητικό ρυθμό. Θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Και γι' αυτό θα παρουσιάσουμε μια πολύ ξεκάθαρη και φιλόδοξη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα το 2030. Και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβεί στι πιο φιλόδοξε ε, δυνατέ δεσμεύσει στην επόμενη ε, διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών για την βιοπικιλότητα των ΗΠΑ στην Κίνα τον επόμενο Οκτώβριο. Και εδώ δηλαδή στο τομέα του κλίματο θα πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο και μπορούμε να το κάνουμε μεταξύ άλλων και στον τομέα, στον κλάδο τη παραγωγή τροφίμων. Και εδώ θα υπάρξει και σχετική πρωτοβουλία τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία από το αγρόκτημα στο πιάτο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα. Οι πυρκαγιέ, για παράδειγμα, στον Αμαζόνιο αλλά και στα διάφορα παρθένα ζά στην Κεντρική Αφρική και στην Νοτανατολική Ασία έχουν καταδείξει το πόσο επίγον είναι να προστατεύσουμε τα δάση μα. Κανένα δηλαδή δεν μπορεί να πει τη σήμερα ημέρα στου ε, διεθνού μα εταίρου ότι δεν μα αφορά αυτό. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με παγκόσμιου πόρου. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να δακτυλοδεικτούμε του άλλου όταν δεν κάνουμε πολλά από τη δική μα πλευρά. Άρα λοιπόν μπορώ να σας παρουσιάσω την επόμενη ιδέα. Ε, τα ε, ε, δέντρα καθαρίζουν τους, ε, τον αέρα μας, ε, ψυχραίνουν τις πόλεις, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και γενικά μας κάνουν όλους να νιώθουν καλύτερα. Άρα λοιπόν ας ξεκινήσουμε ένα τεράστιο project αναδάσωση στην Ευρώπη. Ας αποκαταστήσουμε τα δάση μα και α έχουμε περισσότερε πράσινε περιοχέ μέσα στι πόλει μα. Α δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σχέδιο έτσι ώστε όλε οι πόλει και όλε οι περιοχέ να έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με του υπόλοιπου ε, τι καλύτερε πρακτικέ που έχουν εφαρμόσει και τι πιο επιτυχεί. Και η Πράσινη Συμφωνία δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τι διασκέψει, τι διεθνεί διασκέψει για τη βιοποικιλότητα κάπου μακριά, αλλά και σε ό,τι αφορά τη ζωή γύρω μα. Και το ε, ωραίο σε αυτό είναι ότι όλοι μπορούν να συμμετάσχουν ε, βλέποντα δηλαδή το απτό αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουν. Και επίση θα πρέπει να αποβεί προ όφελο τη υγεία το Green Deal των πολιτών μα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί προ ένα περιβάλλον με μηδενικέ εκπομπέ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντο, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και των ε, υδάτων, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των χημικών, ε, των βιομηχανικών εκπομπών, των φυτοφαρμάκων, των ενδοκρινικών διαταρακτών, των μικροπλαστικών. Ε, για παράδειγμα, τα ε, μικροπλαστικά είναι από του μεγαλύτερου δολοφόνου εντό εισαγωγικών στην Ευρώπη. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ε, ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση ευθύνεται για 400.000 πρόωρου θανάτου στην Ευρώπη ετησίω. Πώ μπορούμε να το αποδεχτούμε λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον πλανήτη μα και θα πρέπει να περάσει η κυκλική οικονομία στο επόμενο επίπεδο. με την πρόληψη δηλαδή τη δημιουργία περισσότερων απορρίμματων. Θα πρέπει να μειώσουμε τα απορρίμματα, να επαναχρησιμοποιούμε και να κυκλώνουμε τα υλικά που έχουμε, έτσι ώστε να έχουμε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Θα σας προτείνω ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που θα εστιάζει στα βιώσιμα ε, προϊόντα και στην χρήση των πόρων, ειδικότερα σε τομείς οι οποίοι έχουν ε, ιδιαίτερα ενεργοφόρα βιομηχανία όπως η κλωστοβιβαντουργία και ο οικοδομικός κλάδος. Αξίτημα μέλη, οι μεταφορέ είναι ένα από του πιο υπογόνου τομέ. Ε, παντού στην Ευρώπη οι άνθρωποι εξαρτώνται από το οχήματά του ε, για την ποιότητα τη καθημερινή του ζωή και ε, συχνά και για την διαβίωσή του. Το γνωρίζω αυτό και δεν θέλω μια Ευρώπη χωρί αυτοκίνητα. Θέλω αυτοκίνητα χωρί εκπομπέ και θέλω οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική μεταφορά. Πρέπει να μειώσουμε τι εκπομπέ και στι αεροπορικέ μεταφορέ και στον ναυτιλιακό τομέα, εάν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε του στόχου για το κλίμα. Αυτό σημαίνει σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα χρήσιμο μείγμα εργαλείων. Πρέπει να επενδύσουμε, για παράδειγμα, στι ε, σιδηροδρόμου. Γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν να περιστούν περισσότερο χρόνο σε ένα αεροδρόμιο, να περιμένουν για πτήση και όχι να είναι σε ένα τρένο για να φτάσουν στον προορισμό του. Αυτό είναι γιατί είναι φτηνότερο. Εμεί χρεώνουμε την πιστοτική κρίση τη ε, κάρτα τη μάνα γη ε, και δεν έχει την πολυτέλεια να το πληρώσει. Θα πρέπει λοιπόν να μην το θεωρήσουμε απειλή για τον τομέα των μεταφορών. Είναι μια προσφορά και θέλω να ενδυναμώσω τον τομέα, να υπάρχουν καθαρά, αποτελεσματικά και προσιτά ω προ την τιμή οχήματα και υποδομέ. Θέλω η Ευρώπη να έχει το καλύτερο σύστημα μεταφορών στον κόσμο. Το, η Πράσινη Συμφωνία θα επιτύχει μόνο εάν όλοι οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν. Εάν πραγματικά έχουμε λοιπόν το Green Deal κοντά μα, στα σπίτια μα στην ουσία. Για να φτάσει αυτό στου ανθρώπου, πρέπει η Συμφωνία για το Κλίμα να αποτελέσει ακρογωνια λίχθο του Green Deal. Η Συμφωνία για το Κλίμα θα συγκεντρώσει πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις από κοινότητες, επιχειρήσεις και γειτονιές. Ανταλλαγή δεδομένων και ε, γνώσεων, έμπνευση για, για τους όλους και καλύτερες πρακτικές και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δείτε τι καταφέραμε να έχουμε με την ε, πρωτοβουλία αυτή τη φορά ε, ψηφίζω και τη σχετική εκστρατεία. Τι έκανε η Επιτροπή των Περιφερειών, ε, τις πρωτοβουλίες δημάρχων σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε τι κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά κυρίως κοιτάξτε τι κάνουν τα παιδιά μας. Δημιουργούν ένα παγκόσμιο κίνημα ε, για να βοηθήσουν τον κόσμο να γίνει καλύτερο. Όλοι μπορεί να είναι το καλό παράδειγμα. Οι καλέ επιλογέ ε, εμπνέουν και ε, οδηγούν σε μίμηση. Δεν υπάρχει υψηλότερο πράγμα από το να εμπνέουν τα ίδια του τα παιδιά, θεωρώ. Αγαπητοί φίλοι, ε, μίλησα κυρίω για το τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Αλλά ε, κυρίω υπάρχει μια τεράστια διεθνή διάσταση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε του άλλου για να αυξήσουν και αυτοί τι φιλοδοξίε του. Είμαι απόλυτα ε, δεσμευμένο ε, στην ενίσχυση τη διεθνή κλιματική διπλωματία και την εφαρμογή των βιώσιμων στόχων. Με τον Green Deal η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει το καλό παράδειγμα, αλλά θα πρέπει επίση να είμαστε προετοιμασμένοι να σκεφτούμε και άλλα μέσα. Για παράδειγμα, ένα φόρο ε, συνόρων για τον άνθρακα, για να έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, εάν οι άλλες χώρες δεν κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς. Ως οικονομικός γίγαντας έχουμε τεράστια μόχλευση για τις εμπορικές μας σχέσεις. Μπορούμε να θέσουμε λοιπόν παγκόσμια πρότυπα και να χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευσή μας όσο καλύτερα μπορούμε για να πείσουμε ότι εν τέλει μπορούμε να είμαστε όλοι και να ζούμε όλοι καλύτερα. Αξιότιμα μόλι και αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο, αλλά πρέπει να επιτύχουμε και βραχυπρόθεσμα κίνητρα. Επίση, πρέπει να βοηθήσουμε και του ανθρώπου που ανησυχούν πώ θα τα βγάλουν πέρα στο τέλο του μήνα. Οι αλλαγέ που απαιτούνται είναι χωρί προηγούμενο και απαιτούν συνεργασία, αποφασιστικότητα και φυσικά και ευφυα. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο. Ποτέ δεν έχω δει κάτι στην Ευρώπη που να είναι εύκολο τουλάχιστον κάτι που να αξίζει τον κόπο. Τα πάντα, ό,τι αξίζει τον κόπο, είναι ε, περίπλοκο. Αλλά γι' αυτό αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Αν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν θα χρειαζόμασταν κοινοβούλιο, δεν θα χρειαζόμασταν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώ είναι περίπλοκο, επειδή είναι περίπλοκο πρέπει να το κάνουμε, αλλά και γιατί είναι το σωστό. Βρίσκομαι εδώ ενώπιον σα ω φίλο και εταίρο, ε, διατεθειμένο να απαντήσω στι ερωτήσει, να συνεργαστώ μαζί σα για να δικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Να το κάνουμε για του ανθρώπου που μα έφεραν εδώ, του Ευρωπαίου πολίτε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ε, με τον πρώτο γύρο ε, ερωταπαντήσεων με τους συντονιστές. Ε. το ΕΛΚ έχουμε την κυρία Στρεντιλάνγκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και καλώς ορίσατε, Φρανς Τιμερμάντσε. Είδαμε και ακούσαμε ένα τμήμα των εντυπωσιακών γλωσσικών σα ικανοτήτων σήμερα. Για να αυτό θα προχωρήσω και θα κάνω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά για να ακούσουμε κι άλλα. Στη γραπτή σα απάντηση αναφέρεται ότι με την γενιά των πατέρων μα και των ε, παππούδων μα ε, ζήσαμε και την ενεργειακή μετάβαση ε, για τα ανθρακοριχεία που κλείσαν στο Λιμπούργο. Και εγώ από το Γέρλε ήμουν και ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή ε, είχαμε έντονα προβλήματα και ακόμα ενδεχομένω, έχουμε και πολλοί ανησυχούν λοιπόν στην περιοχή αυτή γιατί θέλουν να συμβάλλουν αυτό από τη αναλογία αλλά θέλουν να μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους στην τελική ανάλυση. Και βασικά έχει προβλήματα και η βιομηχανία. Και εδώ θα επικεντρωθώ για το ΕΛΚ. Μια φιλόδοξη πολιτική θα πρέπει να προσπίσει και τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα. Την ε, καθαρή βιομηχανία, συχνά καθαρή βιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν και κλιματική πολιτική, να υπάρχει και βιομηχανική πολιτική. Ερωτώ λοιπόν πώ θα συνεργαστείτε με τον Αντιπρόεδρο Βέσταγκερ και με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη που είναι υπεύθυνο για θέματα βιομηχανικής πολιτικής ακριβώς για να πετύχετε τη συνεργασία αυτή, τη συνέργεια αυτή. χαίρομαι που μπορώ να απαντήσω και στα Ολλανδικά. Και όντω ε, είμαι από περιοχή ανθρακορίχων ε, και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν ανθρακορίχοι. Και η πόλη του Χέρλε ήταν η, πιο, η δεύτερη πιο πλούσια πόλη της Ολλανδίας. Σε 50 χρόνια μετά από το κλείσιμο των ανθρακοριχείων είμαστε μία από τις πέντε πιο φτωχές πόλεις ε, της Ολλανδίας. Δηλαδή, ακόμα και σε μια χώρα η οποία είναι πάμπλουτη όπως η Ολλανδία, μια τέτοια μετάβαση σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ομαλή. Κοιτώντας, λοιπόν τι γίνεται στη Γαλλικία, τι γίνεται στην Σιλεσία, περιοχές στην Ελλάδα, στη Γερμανία, όπου υπάρχει ακόμα εξάρτηση από τον άνθρακα και ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, και σκέφτομαι τη δική μας ιστορία, ε, έχω να σας πω μην το παίρνετε στα ελαφριά αυτό. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση και μάλιστα το θεωρούν ε, τόσο μεγάλη πρόκληση που δεν θέλουν να γυρίσουν σελίδα. Γι' αυτό λοιπόν ως Ευρωπαίοι έχουμε τεράστιο καθήκον να βοηθήσουμε και να συνοδεύσουμε τις περιοχές αυτές για να περάσουν σε μια νέα οικονομία, να δημιουργηθεί μια νέα οικονομία. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να σχηματίσουν νέες οικονομίες. Και εκεί λοιπόν χρειάζομαι και την κυρία Φεστάγκερ και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στους συναδέλφου. μου, για μια οικονομία και μια στρατηγική η οποία θα είναι κοντά στην αγορά. Θα είναι σωστή χρηματοδότηση ε, με το σχέδιο Juncker, αλλά να, να χρηματοδοτήσουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι στην αγορά. Για παράδειγμα, η κατάρτιση των πρώην ανθρακορίχων. Αυτό δεν θα το πληρώσει η αγορά. Θα πρέπει εμεί με τα χρήματα των προηγουμένων να το προβλέψουμε αυτό. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έναν ομοιογενή και συνεκτικό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν όλοι σπρώξουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Γεωργία, βιομηχανία, άνθρακα, αλλά και για όλες τις άλλες βιομηχανίες οι οποίες θα πρέπει να περάσουν ε, από μετάβαση. Και αυτό δεν μπορώ να το πετύχω μόνος μου παρά μόνο με τη βοήθεια των συναδέλφων. Ε, επερώτηση να πούμε και κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί αναφερθήκατε ε, στην Σιλσία, στην Πολωνία και στην περιοχή κλείνουν ανθρακοριχεία ε, και θα χαθούν τα επόμενα χρόνια 15.000 θέσεις εργασίας. Και ξέρουμε ε, στην Ευρώπη που θα υπάρξουν τα προβλήματα στην Ισπανία, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι οι χώρες αυτές ε, λένε ότι κοιτάξτε, αυτές οι θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να διασφαλιστούν, να εξασφαλιστούν με κάποιο τρόπο, με μια κατάρτιση για να προετοιμαστούμε ε, με τη μετάβαση αυτή, ακόμα για αυτό το αμοιωτική μετάβαση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε από χρηματοδοτική άποψη τον κόσμο αυτό. Θα χρειαστούμε παραπάνω μέτρα. σω ε, λιγότερο ακτιβισμό από τη Δυτική Ευρώπη και πιο πολύ οικοδόμηση γεφυρών. Πώ θα τι πείσουμε λοιπόν αυτέ τι χώρε πέρα από το Ταμείο Μετάβαση. Ε, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τους Πολωνούς. Απάντηση. Εμάς, δικός μας καθήκον θα ήταν στην Πολωνία, στην Ελλάδα, στη Σλοβακία, στην Ισπανία, σε ένα τμήμα της Γερμανίας, σε πολλά κράτη-μέλη, όπου ξέρουμε ότι θα πρέπει να εγκαταλείξουμε αργά ή γρήγορα τον άνθρακα, να δώσουμε λοιπόν μια εναλλακτική προοπτική στις περιφερειές αυτές, η οποία θα δείξει πώς μπορούμε να κινηθούμε προς μια νέα οικονομία κούτσα στραβά. Η αγορά εργασία στην Πολωνία και στη Σλοβακία είναι πολύ ε, ευίων. Όχι όμως στις περιοχές οι οποίες πλήττονται. Άρα είναι εύκολο να λέμε ότι, α, ξέρετε, θα έχετε κάπου αλλού θέσεις απασχόλησης. Η περιοχή αυτή όμως τι θα κάνει. Αν θέλουμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει στη νέα κυκλική οικονομία να δώσουμε μια εναλλακτική προοπτική στις περιοχές αυτές. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με το InvestEU, το έχουμε πετύχει και θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι πόροι που έχουμε στην Ευρώπη να μπουν στο μηχανισμό για την δικαίη μετάβαση, προκειμένου όλοι οι πόροι να στοχοθετηθούν, να μπουν στην υπηρεσία των περιοχών αυτών. Πολλά χρήματα λοιπόν μπορούμε να εκνοποιήσουμε και ιδιωτικού πόρου, εθνικού πόρου, ευρωπαϊκού πόρου. Στη συζήτηση που θα προκύψει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να πείσουμε και τι δύο πλευρέ ότι είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί η Ευρώπη για την νέα αυτή οικονομία και από πλευρά ε, του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Κύριε Τίμερμαν, παρακαλώ να τηρείτε το ένα λεπτό που έχετε για τι απαντήσει λέει ο πρόεδρο. Από σοσιαλιστέ και δημοκράτε Γκουντιράντ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε υποψήφια εκτελεστική αντιπρόεδρε, θα μιλήσω Σουηδικά και θα ήθελα να δω αν θα μου απαντήσετε στα Σουηδικά. Πάντα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα βρουν εσά στο τιμόνι για την πράσινη αυτή συμφωνία, μία από τις πιο σημαντικές μεταβάσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα στο έργο αυτό να είσαστε η Γκρέτα Τούνμπερκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ε, οι πολίτες και κυρίως οι νέοι που ε, ξεκινούνται στους δρόμους για το κλίμα απαιτούν να λάβει συγκεκριμένη δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζονται για να τηρήσουμε τον στόχο του 1,5%. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε αυτή την κλιματική ουδετερότητα και να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μέχρι το 2030, αν θέλουμε να έχουμε την παραμικρή ελπίδα. Σε αυτούς τους πολιτικούς λοιπόν στόχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία προσέγγιση δύο επιπέδων σε ό,τι αφορά τους στόχους του 2030. Και αυτό προκαλεί ανησυχίες και από πολιτική άποψη, αλλά και από πρακτική άποψη. Πείτε μας λοιπόν, θα αποδεχτείτε αυτή την πρόκληση μέσα σε 100 ημέρες να υποβάλλετε ένα νομοσχέδιο για να αυξηθούν οι στόχοι για το 2030 σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 50%. Εκτός μικροφώνου. Our arguments will be more convincing. Τα επιχειρήματά μα θα είναι πιο πιστικά αν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Ε, για μένα δηλαδή θα αποτελούσε τεράστια έκπληξη το να οδηγηθούμε σε οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα βάσει αυτά τα δεδομένα ότι χρειαζόμαστε κάποια μείωση ε, χαμηλότερα από 55%. Αλλά βέβαια θα είναι, μπορεί να είναι πιο ε, εύκολα υποστηρίξιμη με δική μου θέση αν έχουμε και την απαραίτητη επιστημονική ανάλυση. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ω Επιτροπή 50% και κατά προτίμηση 55%. Αλλά ας κάνουμε και την απαραίτητη έρευνα. Αλλά βέβαια σας ξαναλέω, θα αποτελούσε τεράστια έκπληξη για μένα εάν προταθεί κάτι άλλο, δηλαδή χαμηλότερο το 55% στο 2030. Και αυτό ε, ε, προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε με το μακροπρόθεσμο στόχο του 2050 και μετά έχουμε όλο και περισσότερα εγκύτερα προ εμά. Και βλέπουμε ποια είναι τα ορόσημα. Δηλαδή, μέχρι πότε πρέπει να έχουμε φτάσει σε ποια καμπή, ε, έτσι ώστε να, έχουμε, να χαρτογραφήσουμε αν θέλετε την πορεία στο 2050. Δηλαδή ε, δεν μας επαρκεί μόνο να λέμε μέχρι το 2050 τι θα πρέπει να έχουμε πετύχει, θα πρέπει να ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε, ε, να έχουμε κάνει αύριο, σε δύο χρόνια από τώρα και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Πότε λοιπόν θα έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα επιστημονικά δεδομένα που θα υποστηρίξουν ακριβώ την απόφαση που θέλετε να λάβετε ω Επιτροπή. Και υπάρχει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό ε, ερώτημα που θα ήθελα να θέσω και αφορά του καταναλωτέ μα, οι οποίοι θέλουν να λαμβάνουν ενημερωμένε αποφάσει και οι οποίοι γνωρίζουν ε, πολύ καλά ε, ποιο είναι και ο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή των επιλογών του. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα προϊόντα τα οποία παράγονται τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκείνα που εισάγονται έξωθεν. Έχουμε δηλαδή πρόσφατα πω οι απαιτήσει των καταναλωτών μα έχουν οδηγήσει της ε, παγκόσμιας αλυσίδας ε, λιανικής να παράγουν με λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλλουμε δηλαδή τέτοιου είδους απαιτήσει και στα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο εκείνα τα οποία παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να το εφαρμόσουν αυτό σε όλη την αλυσίδα της παραγωγή αξία. Απάντηση. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα αντίκτυπο στην, στο παγκόσμια, θα πρέπει να έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μα ε, πριν από τη Γλασκόβη, όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, ε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πάμε στη Γλασκόβη και να πούμε ε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρο τη ερώτησή σα, ε, ναι, ε, οι πολίτε μα θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και. Ε, και ο λόγο για τον οποίο καταφέραμε πολύ γρήγορα να περάσουμε και την κατάλληλη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα πλαστικά ήταν ακριβώ επειδή υπήρξε και αυτή η πολύ αποφασιστική στάση από την πλευρά των καταναλωτών μα. Και γνωρίζω πω οι καταναλωτέ μα θέλουν να γνωρίζουν ότι τα όσα έχουν στο τραπέζι του ω τρόφιμα, για παράδειγμα, δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν συμβάνει στην αποψήλωση των δασών. Θα πρέπει να είμαστε θέση να πούμε στου καταναλωτέ μα ότι τα λόγω προϊόντα, τα λόγω τρόφιμα δεν σχετίζονται με περιπτώσει τέτοια αποψήλωση. Αλλά σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και θα πρέπει να συνεργαστούμε με του διεθνεί μα εταίρου έτσι ώστε να το επιτύχουμε. Γιατί ακριβώ το 80% τη ε, αποψήλωση παγκοσμίω που λαμβάνει η χώρα είναι ακριβώ αποτέλεσμα τη αναζήτηση νέων καλλιεργήσιμων εδάφων. Και αυτό ε, βέβαια μπορεί να έχει ω αντίκτυπο ε, και να επηρεάζει και τα τρόφιμα τα οποία έχουμε στο τραπέζι μα, αλλά και τι ζωοτροφέ που χρησιμοποιούμε στην κοινοτροφία μα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί σε σχέση με αυτό και προσεκτικοί. Για το Renew, ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίσετε και σε κάτι το οποίο θα έχουμε αύριο ως ε, πηχαίο τίτλο σε εφημερίδες. Καλωσορίσατε στο σοου του Πραν Τίμερμανς και θα χτυπούνε και τα τύμπανα από πίσω. Ε, Μία συζήτηση που έγινε για το ένα καναφθαρό πλανήτη για όλου. Οι πληροφορίε που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε ότι όλε οι βασικέ αλλαγέ θα πρέπει να υλοποιηθούν από το 2030 και μετά. Μέχρι τότε όμω, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε ενταχθεί σε μια νέα κατάσταση. Πώ βλέπετε λοιπόν να προχωρούν τα πράγματα, Θα προτιμούσατε να διαγράψετε τι προηγούμενε αποφάσει για το σύστημα εμπορία τη εκπομπή ε, το Σιέφ για την ε, χρήση των γεών, ε, τα ε, θέματα της κλιματικής αλλαγής και να κρατήσετε τους στόχους για το κλίμα των Παρισίων και να ξεκινήσετε αμέσω μια αξιολόγηση επιπτώσεων ή θα προτιμούσατε να περιμένετε αυτό το παράθυρο του 2030 και να ξεκινήσετε μια πορεία με μια απαραίτητη 10% γραμμική μείωση η οποία θα ανταποκρίνεται σε αλλαγές ε, και θα έχουμε και αντίστοιχε αλλαγέ ε, στην νομοθεσία. Στην πρώτη περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα θα σα επικρίνουν γιατί έχετε νομοθεσία η οποία είναι ασύνδετη και δεν επιτρέπεται τι επιχειρήσει ε, να σχεδιάσουν τι επενδύσει του. Και στη δεύτερη περίπτωση θα σα επικρίνουν γιατί δεν θα μπορέσετε να διαβάσετε αυτό που γράφει στου τοίχου με πολύ μεγάλα γράμματα. Ποια οδό θα επιλέξετε εσεί λοιπόν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ του ενό ή του άλλου. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα μείγμα των δύο. Πρέπει να επεκτείνουμε το σύστημα εμπορία εκπομπών και σε άλλου τομεί, όπως για παράδειγμα τι αεροπορικέ μεταφορές και στην αυτιλία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και στην κείμενη νομοθεσία η δυνατότητα να... Ε, ε, βρούμε και πιο σκληρά πράγματα για τις εκπομπές, μπορεί να ανανεώσουμε και τις οδηγίες για την ενέργεια και άλλες οδηγίες. Πολλές οδηγίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των δύο. Πάντα θα έχουμε ένα αμάλγαμα πολιτικής μεταξύ των δύο. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο και σε κάποιου τομεί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω παρεπιπτόντω ότι η βιομηχανία έχει αφυπνιστεί και αντιλαμβάνεται παγκοσμίω ότι θα πρέπει να γίνουν πιο σκληρά τα πράγματα και ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν ακόμα και πιο αυστηροί κανόνες. Ε, το IPCC σαφώς μας κατευθύνει προς αυτή την οδό αν ε, δεν θέλουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία του, του πλανήτη το πολύ μέχρι 1,5 βαθμό Κελσίου. Θα, ορισμένες φορές αυτό σημαίνει ότι θα τροποποιήσουμε την κείμενη νομοθεσία, ορισμένες φορές σημαίνει ότι θα νομοθετήσουμε εκ νέου και με τη βοήθειά σας αυτό είναι σαφές. Έχω δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και το Συμβούλιο, να είναι σε θέση να κινηθούν πάρα πολύ πολύ γρήγορα, εάν το επιθυμεί το ευρύ κοινό και υπάρχει και η αίσθηση του κατεπήγοντος. Επομένως αυτό δεν με ανησυχεί καθόλου. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Σίγουρα βεβαίω η πρόκληση θα είναι να υπάρχει κατάλληλο προπολογισμό. Και χάνετε το μικρόφωνο του ομιλητή. Μήπως μπορείτε να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κάποιος μου έσβησε το μικρόφωνο. Χρειαζόμαστε περίπου 200 δις ετησίως για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Τα κράτη-μέλη είναι το ίδιο σφιχτά όπως ε, και οι Ολλανδοί. Γιατί πρέπει λοιπόν να κάνετε κάτι για να τους πείσετε να πληρώσουν, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρήματα για να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Φυσικά. Είδα όμω και μια επιστολή την οποία υπογράφει και ο Ολλανδό Υπουργό ότι πρέπει να φτάσουμε στο μείον 55% μέχρι το 2030, την οποία υπογράφουν και πολλοί άλλοι υπουργοί. Υπάρχει λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντο και στου κάτω χώρες, ε, ναι, η χώρα εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά τι θα ξοδέψει. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε μια πρόταση επιτάπητο ε, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα λέει ότι ναι, μεν φαίνεται να είναι λίγο παραπάνω από αυτό που θέλετε να ξοδέψετε, από το 1,000, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία πολύ πιο γρήγορα και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν οι πολίτες και η βιομηχανία θα πρέπει να αλλάξει και αυτό να αποτελεί δέλεαρ. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δεχτούν αρκετές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου, ελπίζω. Σας ευχαριστώ και άλλη μία λοιπόν Ολλανδική Πρωτοκία από τον Μπάς Άικχοτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από πίσω, κύριε Τίμερμαντσε, και καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σα και για τα λόγια σα που μα ανέπνευσαν για την πράσινη αυτή συμφωνία. Αλλά παρόλα αυτά, να εστιαστούμε λίγο παραπάνω για το κλίμα και τι μπορούμε να περιμένουμε για το χρόνο. Γιατί το χρόνο ήταν η κατεξοχήν χρονιά που θα πρέπει να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Τα τελευταία χρονιά, πρωτού ε, ξεκινήσει επίσημα το Παρίσι. Και είπατε ότι δεν θα σα προκαλέσει έκπληξη το γεγονό αν είμαστε στο μείον 55% από, την ανάλυση, από τις αναλύσεις. Αυτό ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχει μια προσέγγιση δύο επίπεδων, γιατί ήταν λίγο σαφέ από τι απαντήσει σα, τι γραπτέ απαντήσει σα. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε τη μία προσέγγιση 50% και 55%. Έχουν γίνει πολλέ αναλύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη είναι στο δρόμο για το μείον 46%. Κοιτώντα την κατάργηση σταδιακή του άνθρακα κτλ., είμαστε στο μείον 50%. Όλε λοιπόν οι έρευνε μα καταδεικνύουν ότι το 50% θα το πετύχουμε business as usual, αν αλλάξει τίποτα. Άρα αυτό που μα λέτε τώρα θα είμαστε στο μείον 55% όταν θα υποβάλλετε την προτάση σας για την νομοσχέδια για το κλίμα. Μπορούμε λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να υπάρχει λίγο σαφήνεια για το τι συζητάμε. Απάντηση. Μπας. Ο γνωστός μπας. Φανταστική ερώτηση. Κοιτάξτε, η θέση δική μου είναι η εξής. Συμφωνώ μαζί σας Λέτε ότι δεν έχουμε χρόνο για να έχουμε μια δετή προσέγγιση. Ελπίζω όμως και λέω το εξή ότι να πάμε, για να πάμε από το 45% στο 50% έως το 55%, ιδιαίτερα από το 50% στο 55%, θα σημαίνει πολύ σκληρά επιπλέον μέτρα. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να μελετήσει καταρχάς την εφικτότητα αυτού. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό είπε και η Ursula von der μπροστά στο κοινοβούλιο σα. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα επαναλάβω το εξή. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια θέση η οποία να μπορεί να υπάρχει, να, να και σε διεθνέ επίπεδο. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και θα το πω και πριν τη Γλασκόβη στη συνάντηση ΚΟΠ του χρόνου. Αυτή θα είναι η πορεία μου. Μπα και νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρο και επαναλαμβάνω ότι θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η έκπληξη αν καταλήξουμε σε οποιοδήποτε διαφορετικό αποτέλεσμα, σε ό,τι αφορά το μείον 55%. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πιο πιστικό αν κάνουμε μία ανάλυση για να καταδείξουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ δεν θα επιμείνω για το 2030, αλλά θα επιμείνω για το κλιματικό νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τις 100 ημέρε. Γιατί ω τώρα έχω ακούσει λόγια για την ε, κλιματική ευωτερότητα, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει συμφωνήσει και η φυστάμενη απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε τι πρώτε 100 ημέρε, να σα κάνω μερικέ προτάσει, γιατί έχουν γίνει ήδη αναλύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2040 από τι αναλύσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπομπέ για τι διεθνεί αποστολέ, στι ναυτιλικέ αποστολέ, να έχουν μειωθεί κατά 28% μέχρι το 2040. Στην αεροπορία κατά 20% περικοπή μέχρι τον 2030. Ε, 2050. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι ο τομέας ε, των μεταφορών επιτέλους θα μετακινηθεί και επιτέλους ε, θα πρέπει η αρμοδιότητα να είναι στη Γενική Διεύθυνση για το κλίμα, γιατί αυτό θεωρώ θα διευκολύνει πολλά πράγματα. Απάντηση. Κοιτάξτε, για να είμαι εντελώ ξεκάθαρο, να πω το εξή, ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα σε πολλού τομεί, συμπεριλαμβανομένου και του ναυτιλιακού και αεροπορικού κλάδου. Δεν ξέρω, μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό και αργότερα. Κατά δεύτερον, αυτό θα χρειαστεί να το μελετήσουμε. Πόσα μπορούμε να βάλουμε σε μια περιβαλλοντική νομοθεσία, γιατί αφενός δεν θέλουμε να είναι κενή σημασία να λέμε «Α, κοιτάξτε, τότε στόχος με το 2050». Από την άλλη, πρέπει να δούμε και πόσο περιθώριο λιγμού θα δώσουμε στα κράτη-μέλη για να επιλέξουν το σωστό αμάλγαμα βάση και των εθνικών σχεδίων δράσης Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο. Και αυτή τη διαδικασία λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε τώρα. Τα σήματα είναι σαφή, μας τα δίνετε, μας βοηθάτε στη διαδικασία αυτή. Αλλά θέλω να έρθω ενώπιον του Κοινοβουλίου με ένα σχέδιο νομοθετήματο, το οποίο θα πάει αρκετά μακριά και θα διευκρινίζει όχι μόνο που θέλουμε να είμαστε το 2050, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε στον διάμεσα βήματα για να το πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Σαρντόνε από το ID. Καλησπέρα σας. Κύριε Τίμερμανς, η επιτροπή αυτή φαίνεται ότι κρέμεται από τα χείλη της Γκρέτα Τούμπεργκ, αλλά δυστυχώς ε, φαίνεστε σαν πολλούς από τους μαθητές που πηγαίνουν στις διαδηλώσεις για το κλέμα και δεν γνωρίζουν πολύ καλά για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί. Δηλώσατε ότι έχετε ως προτεραιότητα το κλίμα και ξεχάσετε τελείως την υγεία και την διατροφική ασφάλεια. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι σημαίνει να έχουμε κλιματική οδετερότητα το 2050 με ένα κόσμο ο οποίος ε, δεν εκπέμπει καθόλου αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου σε μόνο 30 χρόνια. Το έκανε το περιοδικό Forbes για σας και να σας δώσω κάποια στοιχεία. Για να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές ε, πρέπει να μειώσουμε περίπου μεγατόνους πετρελαίου για συναπτά έτη. Όσον αφορά τι απαιτήσει ενέργεια τα επόμενα χρόνια, φτάνουμε στο 1,6 μεγατόνου καθημερινά. Σε τι ανταποκρίνεται αυτό. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Κατασκευαστική τριών πυρηνικών σταθμών κάθε δύο μέρε για 31 χρόνια συνεχώ. Ή 5.000 ε, αιωλικά πάρκα κάθε μέρα για 31 χρόνια. Επίση, ο κίνδυνο για το περιβάλλον δεν οφείλεται σίγουρα στην Ευρώπη. Πώς ε, σκοπεύετε να κάνετε κάποια πράγματα για την Κίνα και την Ινδία που αυξήσαν κατά 200 περίπου τις 100 τα τελευταία χρόνια τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Δεν λέτε τίποτα για τις χώρες, για παράδειγμα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Βαλκάνια. Κάποιο πρέπει να ξυπνήσει και εσά και τη φίλη σας την Κρέτα. Δεν φταίει η Ευρώπη. Την ερώτησή σας φαίνεται περισσότερο μια γιγάτη επιχείρηση marketing και εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε ως Επίτροπος, θα διευκρινίσετε τις συνέπειες του Green Deal για στόχους οι οποίοι είναι ανέφικτοι και είναι απλώς ιδεολογικοί. Απάντηση. Όταν είναι ισχνά τα επιχειρήματα, όταν ο κόσμος πραγματικά ε, αναγκάζεται να επιτεθεί σε μία κοπέλα 16 χρονών. ντροπή να βλέπω τα tweet ε, κάποιου ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πιο ισχυρός άνδρας στον κόσμο. Πραγματικά, επονίδιστο. Ένα κορίτσι που κάνει ένα και μόνο πράγμα. Μας λέει, κάντε κάτι, κάντε κάτι τώρα. Η Γκρέτα έχει δίκο. Η Γκρέτα έχει δίκιο. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μας που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση. Και αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε. Τώρα. Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Και να πω και κάτι ακόμα. Μας είπαν εδώ και χρόνια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δείτε λίγο τι γίνεται. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σε τι σημείο είναι πλέον αποδεκτό ότι στοιχίζει πολύ λιγότερο από όσα λέγαμε στο προελθόν. Είμαστε σε θέση λοιπόν να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία. Και εσεί θέλετε να πάτε στην Ιταλία και να εξηγήσετε στου Ιταλού ότι θα πρέπει να μείνουν κάπω οι παραλίε όπω είναι σήμερα. Είναι απαραδεκτό αυτό στην Ιταλία. Θέλετε να πάτε στην Ιταλία και να εξηγήσετε στου νέου που ζουν στι πόλει, ότι θα πεθάνουν πιο νωρί γιατί δεν είναι καλό ο αέρα που αναπνέουν. Όχι. Ακόμα και αν δεν ισχύουν τα επιστημονικά στοιχεία, ακόμα και αν δεν ισχύουν τα επιστημονικά στοιχεία, έχουμε καθήκον για τα παιδιά μας να εξασφαλίσουμε καθαρό περιβάλλον. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. πληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Σας υποτίμησα. Μιλήσατε σαν καλός μαθητής, εσείς ε, κάνατε απλό η προπαγάνδα, αλλά δεν περιμένατε τίποτα καλύτερο. Δεν απαντήσατε στο ελάχιστο στην ερώτησή μου. Είναι πάρα πολύ αδύναμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν για να μιλήσει για το περιβάλλον κρύβεται πίσω από ένα κορίτσι 16 χρονών όπως η Γκρέτα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Θέλω να ξέρω αν το μεγαλύτερο μέρος της ρήπανση από τα πλαστικά προέρχεται από τις ασιατικές χώρες γιατί δεν κάνετε τίποτα ενώπιον του. Ξεκίνησε η έκτη σύνοδο και η, προσοχή επικεντρώθηκε σε θέσεις των πιο φανατικών περιβαλλοντιστών. Σκοπεύετε λοιπόν να συνεχίσετε αυτή τη μη πρόοδο. Θα επιστρέψουμε τι, στα κάρα με τη, στις άμαξες με τα ε, άλογα. Ε, θα μιλάτε μόνο με τα tweet και με το Instagram. Απάντηση. Πραγματικά πιστεύετε ότι τα πλαστικά μπουκάλια στις ε, παραλίες στην Ιταλία είναι από την Κίνα και από την Ινδία. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και έχουμε καθήκον να καθαρίσουμε εμείς το περιβάλλον μας. Και αυτό θα το λέω πεπισμένο. Εγώ θα πάω στην Ιταλία. Θα πάω και θα μιλήσω και με του δικού σα του ψηφοφόρου. Θέλουμε καθαρό περιβάλλον, ναι ή όχι. Αν θέλουμε καθαρό περιβάλλον, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξει και η βιομηχανία. Πρέπει να αλλάξουν και τα αυτοκίνητα. Γιατί να μην έχουμε αυτοκίνητα χωρί εκπομπέ. Αυτό είναι δυνατόν και πρέπει να το κάνουμε. Α το κάνουμε όλοι μαζί. Okay. Ωραία. Για το ECR, Κύριο Αλεξάνδρ Βόντρα. Welcome to the revolution. Ε, να το πούμε έτσι. Ε, δηλαδή βλέπουμε να έχουν ανάψει τα αίματα εδώ και ε, η δυναμική εδώ είναι απίστευτη. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο ή στις αρχές αυτού του έτους ο προηγούμενος επίτροπος δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό ούτε είναι απαραίτητο να μετατρέψουμε τους στόχους του 2030. Μετά, τον Ιούλιο, η κυρία Ούσρα Φοντερ Λάιν δεσμεύτηκε να υποβάλει ένα σχέδιο το οποίο θα αυξήσει αυτούς τους ε, στόχους ε, για το 2030 στο 55% υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Και τώρα σας ασκούνται πιέσεις από διάφορες χώρες έτσι ώστε να δεσμευτείτε χωρίς καμία ιδιαίτερη προϋπόθεση σε αυτόν τον στόχο του 55%. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω ε, τη βαθιά μου ανησυχία για αυτή τη δυναμική την οποία παρατηρούμε. Δηλαδή ανησυχώ ότι αυτή η πράσινη συμφωνία, του Green Deal, ε, θα έχει κόστος υψηλότερο από αυτό το οποίο μπορούν να αντέξουν οι κοινωνίες μας γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με βασικές ανθρώπινες ανάγκες όπως η στέγαση, η θέρμανση, τα τρόφιμα, οι μεταφορές και θα επηρεαστούν αρνητικά. Ε, ειδικότερα οι ε, οικογένειες ε, του μέσου εισοδήματος ε, και ειδικότερα βέβαια οι πιο χαμηλόμιστοι, γιατί θα υπάρξουν και υψηλότερα ε, υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Εσείς λοιπόν ως σοσιαλδημοκράτης θέλετε κάτι τέτοιο στο πλαίσιο των δικών σας αυτών στόχων. Ε, Ποιε είναι ε, οι συγκεκριμένες απαντήσεις που μπορείτε να μου δώσετε. Ακούσαμε κάποια ωραία λόγια από εσά, αλλά ε, θα πρέπει καταρχήν να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο πρώτο αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους όμορφα όνειρο. Καταρχήν να πω, α, κύριε Βόντρα, σας γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό και ε, θα πρέπει να εκφράσω το θαυμασμό μου για αυτά που έκανε όταν ε, υπό το καθεστώ που βρισκόταν η χώρα του και πραγματικά ε, έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο και το σέβαμε πάρα πολύ. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα διαφωνούμε. Ε, και αναφέρθηκα σε αυτό προηγουμένω ε, στα εισαγωγικά μου σχόλια. Για παράδειγμα, σε αυτό των κοινωνικών κατοικιών, τη κοινωνική στέγαση γενικότερα. Δηλαδή, αν βοηθήσουμε του ανθρώπου να μονώσουν τι κατοικίε του και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά όπου αυτό είναι δυνατό ή να κάνουν συμπληρωματικά μέτρα, θα πρέπει να του υποστηρίξουμε αν δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουν μόνο του αυτές τις επενδύσεις. Γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει, οι λογαριασμοί ρεύματο θα είναι πιο φθηνοί και οι εκπομπέ θα είναι χαμηλότερε. Ε, αυτό χρειαζόμαστε. Είστε ε, απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν ε, λάβουμε κάποια συμπληρωματικά μέτρα για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, την προστασία από τον περιβάλλοντο χωρί να εξετάσουμε τη φορολογική πολιτική, τότε ναι, θα υπάρξουν δυσμενεί ε, συνέπειε για του πολίτε μα. Αλλά θα εξετάσουμε και τη φορολογική πολιτική, γιατί νομίζω πω φορολογούμε τα λανθασμένα ε, αντικείμενα. Δηλαδή, ε, εδώ θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και να επιχειρηματολογήσουμε με τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση των φορολογικών συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντικό αντίκτυπο για, τις, ε, για, την, για του μέσου και χαμηλότερου εισοδήματο. Αλλά από την άλλη πλευρά, και το τονίζω αυτό, αν δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν αναλάβουμε δράση, τότε ε, δείτε τι θα συμβεί ε, στο επίπεδο της κλιματική αλλαγή. Ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Δείτε δηλαδή πώ θα προκύψουν συγκρούσει από αυτού του ελληνικού πόρου και ποιο τελικά θα είναι εκείνο που θα πληγεί πρώτο και θα πεθάνει πρώτο, εάν έχουμε χαμηλότερη ποιότητα ε, ζωή ε, στις πόλεις, μα πάντοτε εκείνοι οι πιο εκατότερες κατώτερες ε, ένταξεις. Κύριο Σεβόντρα και πάλι. Ναι, πολύ ωραία λόγια, αλλά θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένα στοιχεία πρωτού αναφερθείτε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να μας πείτε ακριβώς τι θα υπάρξει και σε επίπεδο αποζημιώσεων, γιατί η Ινδία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βραζιλία και ούτω καθεξής ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ε, συμφωνήσουν μαζί μα. Ε, γιατί το να λέτε ότι θα πρέπει να δώσουμε εμεί το καλό παράδειγμα είναι κάτι το θετικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί στην πράξη. Άρα λοιπόν, ε, τι ακριβώ θα γίνει. Είστε για παράδειγμα διατεθειμένοι να κηρύξετε πόλεμο των εισαγωγικών πέραντι σε αυτέ τι ε, χώρε, αν δεν κάνουν κάτι. Απάντηση τα ίδια επιχειρήματα είχαν αναφερθεί όταν είχαμε δημιουργήσει ε, την ενιαία αγορά. Ότι δηλαδή θα είναι υπερβολικά τα πρότυπά μα, θα είμαστε υπερβολικά ακριβοί και κατά συνέπεια ο κόσμο, οι υπόλοιπε χώρε δεν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα μα και ούτω καθεξή. Όμω, ε, τι έγινε τελικά. Οι υπόλοιπε χώρε, ο υπόλοιπο κόσμο θέλει να συμμετέχει εδώ, να είναι σε θέση να εξάγει τα προϊόντα του εδώ σε αυτή την ενιαία αγορά. Και έχουμε ψηλά πρότυπα αλλά φυσικά υπάρχει εδώ με αχίλιο να εάν σε αυτό το σχέδιο εάν δεν μπορούμε να πείσουμε τι άλλε χώρε του κόσμου να ακολουθήσουν το παράδειγμα μα. Ε, αλλά εγώ είμαι πιο αισιόδοξο από εσά. Ναι, ε, σε εμά αντιστοιχεί μόνο το 9% των παγκόσμιων εκπομπών, αλλά έχουμε ε, και πολύ πιστικά επιχειρήματα. Γιατί και, και οι Κινέζοι δεν θέλουν να εξαντληθούν τα έδατα του, δεν θέλουν να έχουν κακή ατμοσφαιρική ε, ποιότητα και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα από την πλευρά των Ηνωμένων ε, Πολιτειών. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να μην συμφωνεί μαζί μας, αλλά μιλήστε με τους δήμους και ε, Θα δείτε ότι συμφωνούν μαζί μας. Ναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνασπισμούς, μπορούμε να πείσουμε τους υπόλοιπους και είμαι πεπισμένος ότι αποτελεί καθήκον μας και σε ηθικό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε όχι μόνο και την καλύτερη προστασία, αλλά και πολιτική σταθερότητα. Γιατί ακριβώ με αυτέ τι εξελίξει, με την έλλειψη των πόρων, θα έχουμε συγκρούσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά του τους σπόρου πόρους ειδικότητα. Ευχαριστώ. Εκεί η Σιλβία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Μέρμανς. Είναι μεγάλη η έκπληξη. Περιμένουμε ακόμα επιστημονικά στοιχεία για να θέσουμε το στόχο του 55% αν θέλουμε να υπάρξει σωστή στοχοθέτηση στη χρηματοδότηση, θα πρέπει να ξέρουμε πώς, θέλει να, πώς θέλουμε να έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον μέχρι το 2030. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν και ζητώ απευθύνω έκκληση για το στόχο του 55%. Ένα δεύτερο θέμα που θα θέλω να θέσω είναι η βιοπικιλότητα. Άκουσα διάφορους υποψηφίους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστώνω ότι δεν έχουν καθόλου καθεσυχαστεί οι ανησυχίε μου για την βιοπικιλότητα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Να έχουμε υπόψη μας ότι αν η βιοπικιλότητα είναι σε καλό επίπεδο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος με καλύτερο τρόπο. Οδεύουμε προς το χείλος του γκρεμού σε ό,τι αφορά την απώλεια των ειδών. Τι θα κάνουμε λοιπόν και πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Είσαι στο πρώτο θέμα για το είπατε. Τι 55% σημειώσαμε αυτά που είπατε και σαφέστατα μάλλον αυτά θα συνάδουν και θα τα επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιοπικιλότητα τώρα είμαστε σε κίνδυνο να χάσουμε ένα εκατομμύριο από τα 8 εκατομμύρια ήδη στον πλανήτη. Η ε, οι γεννήσει, οι υφαλοί πεθαίνουν, το ίμιση έχει καταστραφεί, η αποδάσωση η αποψήλωση, βλέπετε τι κάνει σε ό,τι αφορά επίσης ε, ε, τα φυτοφάρμακα. Είναι πραγματικά κατεπίγουσα η κατάσταση και πραγματικά είμαστε στο χείλος μιας διεθνούς αφύπνισης σε ό,τι αφορά την απώλεια βιοπικιλότητας, όπως πριν από κάποια χρόνια όταν ε, κάναμε τη Συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος. Τα δύο φαινόμενα προφανώς και συνδέονται η αποψήλωση σημαίνει και ότι εξαντλούμε τα αποθέματα άνθρακα τους. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη με εντατικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη διάσκεψη τον Οκτώβριο του χρόνου για να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πρέπει να λάβουμε δράση σε ό,τι αφορά την διάσωση της βιοποικιλότητας και πιστεύω ότι η ανακοίνωση τη Επιτροπή Γιούνκερ για την καταπολέμηση τη αποψήλωση μπορεί να αποτελέσει ένα απόσπαστο τμήμα αυτή, γιατί χρειάζεται πραγματικά ε, να έχουμε διεθνεί εταιρικέ σχέσει, συνεργασίες. Θα πρέπει οι χώρε στι οποίε πλήττονται να είναι τμήμα τη λύση. και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε και εμεί τι ευθύνε μα, Μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τον τρόπο που καταναλώνουμε. Γιατί ο τρόπο που καταναλώνουμε έχει αρνητική, αρνητικό αντικτύπωση στη βιοπικιλότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν το σύστημα όμως ε, συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, αν τα πράγματα παραμένουν ως έχουν, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα τι γίνεται με τις επιδοτήσεις ε, τις σε επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ακόμα έχουν στο επίκεντρο τα ορεικτά κάψιμα. Όχι μόνο μας εμποδίζουν από το να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά λειτουργούν κατά των στόχων μας. Πώς λοιπόν μπορούμε να κινηθούμε προς μία κατάσταση όπου όλοι οι πόροι θα αποσκοπούν την επίτευξη του κοινού αυτού στόχου. Είσαστε ρητεθειμένος να αμφισβητήσετε την ομοφωνία στον τομέα αυτό. Σε κάποιους τομείς, κοιτάξτε η απάντηση, όπως στην αφρολογία, στην ενέργεια, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η συνθήκη για την επωνομαζόμενη Πασαρέλα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μετακίνηση από την απόλυτη ομοφωνία στην ε, πλειοψηφία. Αλλά το πιο βασικό για αυτά που μας λέτε είναι το εξή. Θα έχω την ευθύνη να εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της δεν θα έχει αντικρουόμενες δράσεις. Και αυτό φαντάζομαι θα είναι ό,τι πιο δύσκολο θα έχω να κάνω σε εσωτερικό επίπεδο. Να εξασφαλίσω ότι όλα όσα κάνουμε θα είναι συμβατά με το στόχο της ε, κλιματικής ουδετερότητα μέχρι το 2050 και σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα. Δεν θα μπορούσα να σας πω και να σας ε, εγγυηθώ στην παρούσα φάση ότι έχουμε απαλείψει οποιαδήποτε πιθανότητα αντικρουόμενων πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να σα το πω αυτό. εδώ πέρα και στο Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι σε κάποιε περιπτώσει οι διαφορετικέ επιτροπέ έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όμω ότι από εδώ και πέρα ό,τι κάνουμε θα έχει τον ίδιο στόχο. Να δημιουργήσει μια βιώσιμη κοινωνία που θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Και εδώ θα χρειαστεί θεωρώ να θεωρήσουμε πολλές από τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων τώρα. Ξεκινάμε και πάλι με το ΕΛΚ και τη Ρομπέρτα Μέτσολα. Ευχαριστώ πολύ. Η μείωση των πλαστικών στους ωκεανούς μας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες των πολιτών. Έγινε το πρώτο βήμα ε, για, με την ε, νομοθεσία για την απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης. Τώρα πρέπει να πάμε τι περαιτέρω. Συμφωνώ με αυτά που είπατε προηγουμένως για τα πλαστικά μπουκάλια στις παραλίες, αλλά αυτή τη στιγμή τα ρεύματα έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν τα πλαστικά και μάλιστα σε θάλασσες χωρών που είναι όμορες με τρίτες χώρες και τα πλαστικά υποτίθεται ε, τα οποία είναι προς ανακύκλωση δεν είναι πάντα βιώσιμα και δεν είναι και καλά σχεδιασμένα. Και τελικά δεν κάνουν τίποτα για το περιβάλλον, απλώς αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τα στέλνουμε στην άλλη άκρη του κόσμου απλώς για να επιστραφούν και να γίνει καύση ή να ε, τα χρησιμοποιήσουμε κάπως αλλιώς. Δεσμεύεστε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πιέσει μέσω των κρατών μελών και σε διεθνή φόρα για να μειώσουμε τα πλαστικά. Η, ε, σύντομη απάντηση στην ερώτησή σα είναι ναι, φυσικά. Αλλά θέλω να το πω λίγο πιο αναλυτικά. Μαθαίνουμε συνεχώ πόσο επικίνδυνα, για παράδειγμα, είναι τα μικροπλαστικά. Νομίζω ότι κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα έρευνα μας δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και για την υγεία μας και για το περιβάλλον. Πρέπει να κάνουμε κάτι από αυτού. Πρέπει να κάνουμε κάτι και για τις συσκευασίε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω για απαγόρευση συσκευασιών ή να εξασφαλίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον συσκευασίε που να περιλαμβάνουν πλαστικά μιας χρήσης Πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι φροντίζουμε τα δικά μα τα σκουπίδια. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή κίνηση τη Κίνα να πούνε ότι δεν δεχόμαστε ευρωπαϊκά πλαστικά μια χρήστη πλέον. Τώρα τα εξάγουμε σε άλλε τρίτε χώρε και αυτό θεωρώ ότι είναι πονίδεστο. Πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε. Πρέπει να φροντίσουμε εμεί τα δικά μα τα απόβλητα. Και ο μόνο τρόπο να το κάνουμε είναι να μην έχουμε. Τα καλύτερα απόβλητα είναι τα απόβλητα που δεν διαθέτει. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη ανακύκλωση, αλλά δεν είναι υπέρτατη λύση. Η υπέρτατη λύση είναι να μην χρειάζεται να γιατί δεν το χρησιμοποιήσει ή αν το χρησιμοποιήσει θα το ξαναχρησιμοποιήσει χωρίς να το ανακυκλώσεις. Βασίζομαι λοιπόν στην υποστήριξή σας όταν θα έχουμε προτάσεις επί του ζητήματος. Ευχαριστώ. Τώρα να περάσουμε στην ισότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ε, τελειώνει το fitness ε, ε, check για το περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα και αποδείχθηκε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση δημιουργεί εκατοντάδες εκατομμυρίων χρέη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ανησυχεί τους πολίτες στη χώρα μου, στη Μάλτα, όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση αυξάνεται και δημιουργεί και ε, ανησυχία στις οικογένειες. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τι ε, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αν θα ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση ε, για χώρε οι οποίε δεν συμμορφούνται προ την νομοθεσία. Αυτό όμω είναι η τελευταία κίνηση για κάποιου οι οποίοι ήδη είναι εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρική ρήπανση. Πώ λοιπόν θα εφαρμόσετε την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι απόλυτα σαφή. Οι κανόνε είναι σαφεί και πρέπει να του εφαρμόσουμε στα κράτη-μέλη. Αυτό που κάνει πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να βρει λύση μέσω διαλόγου με τα κράτη-μέλη, αλλά θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Η νομοθεσία χρειάζεται κατεπηγόντω, αλλά δεν εφαρμόζεται σε πολλά κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση τη και να ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση. Και θεωρώ ότι είναι προσωπική μου ευθύνη να εξασφαλίσω ότι όντω θα γίνει κάτι τέτοιο. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε ε, Τίμερμανς, η ε, πρόεδρος Φονταρ είπε ότι θα προτείνει ένα σχέδιο δράση για να αυξήσουμε τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του 2030, αλλά αυτή τη στιγμή ε, ο στόχος δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκοιμίου του ε, ναυτιλιακού τομέα, δηλαδή αυτή τη στιγμή εξαιρείται ακόμα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει ρύθμιση κανονιστική σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα δυναμητήσουμε οποιασδήποτε άλλες προσπάθειες γίνονται από άλλους τομείς για να επιτύχουμε αυτήν την, τις μηδενικές εκπομπές. Τώρα αναφερθήκατε στη δυνατότητα του να υπάρξουν τέτοιου είδου επεριορισμοί ε, και στον αεροπορικό τομέα και τον ναυτιλιακό. Αλλά στι γραπτέ απαντήσει ε, που δώσατε, είπατε ότι ε, θα αναλάβετε δράση με βάση τι προτάσει που θα γίνουν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την επέκταση του συστήματο εμπορία εκπομπών και σε αυτού του τομεί. Σα καλώ να μην περιμένετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση. Είσαστε λοιπόν διατεθειμένο να προτείνετε από την πλευρά τη Επιτροπή στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του συστήματο εμπορίου εκπομπών αυτή η διεύρυνση λοιπόν να αφορά και τον αυτιλιακό τομέα. Ε, και επίση ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για μα. Εσεί λοιπόν ω αρμόδιο ε, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, πώ θα διασφαλίσετε ε, πως η Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα θα έχει την απόλυτη ευθύνη σε ό,τι αφορά την ε, μελλοντική εφαρμογή του συστήματος εκπορίων εκπομπών και τη διεύρυνσή του ακριβώς στον αεροπορικό και τον αυτιλιακό τομέα. Απάντηση. Να είμαι ξεκάθαρος γιατί εδώ, σε αυτό το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, γιατί δεν ξέρω αν το απάντησα ήδη, ναι, εγώ θα είμαι αρμόδιος και θα υπάρχει συναρμοδιότητα από την κίνδυνη της Μεταφορές, αλλά την ε, βασική ευθύνη θα έχει η Γενική Διεθνή Κλίματο. Εγώ λοιπόν αναλαμβάνω προσωπική ευθύνη για αυτό το τομέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ναυτιλιακό τομέα, ναι, το ETS, το σύστημα εμπορία εκπομπών, θα πρέπει να ε, επεκταθεί και εκεί. Αλλά θέλω να έχουμε και άλλου τομεί. Για παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε πράσινα φιλοπεριβαλλοντικού λιμένε δηλαδή ε, και ε, ηλεκτρισμό. Για παράδειγμα, με την που προέρχεται από αλλού. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν ε, κρουαζιερόπλια, για παράδειγμα, τα οποία εισέρχονται σε κάποιου λιμένε, ε, τα επίπεδα ατμοσφαιρική ρήπανση αυξάνονται γιατί ακριβώ η καύση γίνεται με πολύ ε, ε, βλαβερά ε, ε, υλικά, οπότε καύσιμα. Ουσιαστικά λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε και μέτρα σε ό,τι αφορά αυτούς τους, τους Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ποιε ακριβώς είναι οι εκπομπές των πλοίων και πώς αξιοποιούνται με βάση τους κινητήρες, τη ταχύτητα με την οποία κινούνται τα πλοία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάσουμε γιατί δεν μπορούμε να δεχόμαστε τη σήμερα ημέρα να συνεχίζει να εξαιρείται από αυτά τα μέτρα ο ναυτιλιακός τομέα γιατί οι κινητήρες των πλοίων πραγματικά είναι εξαιρετικά ε, ε, έχουν εξαιρετικά υψηλέ εκπομπέ και δεν είναι δίκαιο απέναντι στου άλλου κλάδου το να εξαιρείται ο ναυτιλιακό τομέα. Η κυρία και πάλι. Ε, ναι, δέχομαι την απάντησή σα, ε, γιατί και εγώ κατάγομαι από τη Μάντα και γνωρίζω ακριβώ τι σημαίνει όταν εισέρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο σε ένα λιμένα εκεί. Και γι' αυτό ακριβώ σα ζητώ να αναλάβετε άμεση δράση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην περιμένετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε όμω στην ατμοσφαιρική ρήπανση και υπάρχει και εδώ και ένα ε, σημαντικό τομέα σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ και εδώ αναφέρομαι στι οδικέ μεταφορέ. Ε, μέχρι στιγμή τα πρότυπα σε ό,τι αφορά το τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, είναι εκείνα που έχουν αποδεχθεί τα πιο αποτελεσματικά. Προτείνεται λοιπόν ε, την συμπερίληψη κατά κάποιο τρόπο ε, το, στο ETS των ε, του τομέα των οδικών μεταφορών και τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα πρότυπα των της αυτοκινητοβιομηχανίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την χρήση και βιώσιμα χρησιμοποιούμενων μπαταριών, έτσι ώστε να έχουμε και ένα βιώσιμο κλάδο μεταφορά γενικότερα. Ναι, ε, ουσιαστικά είναι διάφορε ερωτήσει που μου θέσατε μέσα σε μία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόσουμε την ε, νομοθεσία που ισχύει ήδη σήμερα με κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα ε, και νομίζω ε, πω είτε αυτοκίνητο βιομηχανία ε, δεν μπορεί πλέον να βρίσκεται σε μια βολική και άνετη θέση. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που έπρεπε να κάνει στο παρελθόν και τώρα θα είναι υποχρεωμένη να το κάνει και εμεί θα φροντίσουμε να επιβληθεί η νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τώρα του ETS στι οδικέ μεταφορέ, δεν είμαι επί τη αρχή ε, κατά αυτή τη ιδέα ε, και είμαι υπέρ του να περιληφθεί μέσα στο μείγμα των πολιτικών, αλλά δεν νομίζω πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό ως δικαιολογία για να μην επιτύχουμε τους στόχους μας σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Τα πράγματα δηλαδή ε, ε, είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και απλά όταν έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ και να αναγκάζεται ο κλάδο να συμμορφώνεται με αυτέ τι εκπομπέ. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η εφαρμογή του ΙΔΕΣ e δεν μπορεί να αποτελέσει μέρο του ε, μείγματο πολιτικών μα, αλλά λέω ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να μην ανταποκριθούμε στου στόχου. Και κάτι ακόμα. Ε, ο Μάριο Ευκοπίτη ε, στην Επιτροπή Juncker έκανε. Ε, πραγματικά εξαιρετική δουλειά έτσι ώστε ακριβώ να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και στην αυτοκινητομηχανία σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των ε, μπαταριών και προσπαθούμε τώρα να συμπεριλάβουμε ε, την Ευρώπη σε αυτήν την ε, νέα γενιά των μπαταριών όπου δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή πρώτε ύλε οι οποίε είναι πολύ βραβελέ για το περιβάλλον ή οδηγούν σε σύγκρουση αλλού, είναι πολύ δυσέβρετε, χρειάζονται μεγάλου αποθηκευτικού χώρου και ούτω καθεξή. Αλλά ε, η μπαταρία μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να αποτελέσει δηλαδή μια ευρύτερη λύση σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργεια. Για παράδειγμα, το υδρογόνο θα αποτελέσει σίγουρα ένα πολύ σημαντικό τρόπο αποθήκευση ενέργεια ε, στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Να τηρείτε παρακαλώ το χρόνο ομιλία σα. Και έχουμε τώρα λοιπόν και το χρόνο ομιλία και στι συμπληρωματικέ ερωτήσει για το Renew. Ο κύριο ε, Φεντερλέ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Εκτελεστική Αντιπρόεδρε, υποψήφια. Θα μιλήσω μια γλώσσα που δεν τη μιλάτε, τα σουηδικά. Αλλά είμαι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια θα την έχετε κατακτήσει κι αυτή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ισορροπία, έχουμε α, πολλά και μεγάλα καθήκοντα να επιτελέσουμε σε αυτή τη θετετία πολλές ε, εθνικές και εσωτερικές μάλλον και διεθνείς προκλήσεις αν θέλουμε να τηρήσουμε το συνθήκη του Παρισιού. Βλέπουμε με φρίκη τι συμβαίνει στον Αμαζόνιο. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση από πλευρά της Ευρώπης. Ίσως θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε μια απάντηση με κάποια μέσα. Αλλά προφανώς ο τομέα της γεωργίας είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε για να αποτρέψουμε την αποψήλωση του Αμαζονίου. Βλέπουμε όμω αποψήλωση και στα δάση της Ευρώπης. Μακροπρόθεσμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει και σε άλλες χώρες. Από νομοθετικής λοιπόν άποψης πώς μπορούμε να να πετύχουμε αυτή τη χρυσή τομή για να, υπο, να διατηρήσουμε την α, βιοπικιλότητα και την βιώσιμη δασοκομεία. Απάντηση. Μπορεί και να κάνω λάθο να με διορθώσετε, αλλά εξ όσων γνωρίζω, έχουμε πιο πολλά δάση στην Ευρώπη σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, αλλά δεν έχουμε αποψήλωση στην Ευρώπη. Έχουμε πιο πολλά δάση. Δεν φτάνουν ωστόσο. Χρειάζεται πραγματικά μια στρατηγική για την επαναδάσωση. Για την αναδάσωση. για να μην υπάρχει και αντίφαση με άλλου ε, σκόπου. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δάση σε κάποιες περιοχές δεν βοηθούν τον περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναδάσωση. Για να εξασφαλίσουμε επίσης ότι ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στην δασοκομεία θα είναι τμήμα της λύσης, θα συμπεριληφθεί στην πολιτική που θα καταρτήσουμε και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό στην Ευρώπη θα έχουμε και πιο ισχυρά επιχειρήματα για να πείσουμε άτομα εκτός Ευρώπης που αντιμετωπίζουν τις προκλήσει. Κοιτάξτε πόσο ποσοστό του δάσου χάνεται και ακούμε το επιχείρημα ότι 80% ε, των δασών χάνεται και αποψηλώνεται για να δημιουργηθούν καλλιεργήσιμε ε, γέε. Yes. Από τον Αμαζόνιο κάποιο μου έλεγε ότι περίπου 50% του εδάφους που αποψηλώνεται χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Άρα μιλάμε για τεράστια τεράστιες εκτάσεις που χάνονται σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα, την απορροφησία άνθρακα κτλ. Χρειάζεται λοιπόν διεθνή προσέγγιση και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και χώρε οι οποίε συνήθω διστάζουν, γιατί προφανώ βλέπουν κάποια δυνατότητα οικονομική ανάπτυξη και σε κάποιε περιπτώσει θα πρέπει να εξετάσουμε και τι εισαγάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να του πείσουμε να παράγουν άλλα προϊόντα που δεν προαπαιτούν από ψήλωση και να επιμείνουμε στα προϊόντα αυτά. Νόμιζα ότι ο πρόεδρος θα μου έδινε το λόγο για να συνεχίσω. Μάλιστα. Ε, τα τμήματα αυτά για την ενέργεια. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουμε ποια θα είναι η επόμενη φάση στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμα μια ισορροπία και σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα, αλλά και τα απορρίμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να, χρησιμοποιηθούν για ε, παραγωγή ενέργειας. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, για να κινηθούμε προς τις αρνητικές εκπομπές. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο από τον υποψήφιο επίτροπο για τις αρνητικές εκπομπές. Κοιτάξτε, απάντησε. Είναι, θεωρώ δυνατό, αλλά επειδή είναι οργανικό δεν σημαίνει, βιολογικό δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Τα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, έχουν κάνει τεράστια ζημιά τα τελευταία δεκαετία. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς. Τότε θα μπορέσουν να αποτελέσουν επικοδομητικό στοιχείο της ε, λύσεις στην αεροπορία. Θα χρειαστούμε πιο πολλά βιοκαύσιμα για η ηλεκτρική αεροπορία δεν την βλέπω να πραγματοποιείται ε, σύντομα. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τις εκπομπές, χρειάζεται να κάνουμε ένα διαφορετικό μείγμα καυσίμων. Άρα τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς θα μπορούσαν να παίξουν έναν ενδιαφέροντα ρόλο στο όλο μείγμα αυτό. Αλλά να προσέξουμε κειμένου να μην δώσουμε έτσι μια συνολική έγκριση σε οτιδήποτε είναι βιολογικό. Ευχαριστώ τώρα από το ΕΛΚ η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμαντς. Πανέρχομαι λίγο στις γραπτές, ε, στα γραπτά σχόλια που κάνατε ε, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα. Γιατί δεν αναφερθήκατε σε αυτόν τώρα στην εισαγωγή σας. Αναφέρεστε στην ε, πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά όπως ονομάζεται από το αγρόκτημα στο πιάτο σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Και θα ήθελα να σας θέσω ένα ε, ερώτημα ε, σε ό,τι αφορά αυτές τις πολιτικές. Ε, ε με ενδιαφέρουν πολύ τα σχόλια που κάνατε σε ό,τι αφορά ε, τις που έχουμε στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν τέτοιου είδου αντιφάσει σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη φορά τα τρόφιμα, το εμπόριο και το καθεξή. και, σε ό,τι αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού, αυτό που έχω πει επανειλημμένα είναι ότι ε, δεν ε, προβλέπει τίποτα σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά τα οποία ε, σωματώνονται, αν θέλετε, μέσα σε αυτά τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Δηλαδή, είναι φτηνά τα τρόφιμα με βάση ακριβώ τέτοιου είδου αυτά τα αγαθά, αν θέλετε. Οπότε, πόσο αποτελεσματικό θα είσαι σε σχέση με αυτό. Απάντηση. Ναι, ο χρόνο θα το δείξει, αλλά να απαντήσω και να πω ότι λόγω της επαγγελματική μου εμπειρίας από την ε, δεκαετία του 1980, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 1980 με δραστήριο σε αυτόν τον τομέα της αγροτικής πολιτικής και αυτό που ε, παρατηρώ ξανά και ξανά είναι ότι οι αγρότες οι οποίοι υποφέρουν χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για να προστατευτούν οι πολιτικές που επιθυμούν εκείνοι οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το φαινόμενο. Ε, και νομίζω πως ε, η νέα πολιτική την οποία έχει ξεκινήσει ο Φιλ Χόγκαν αυτή, δηλαδή ε, η νέα λογική σε ό,τι αφορά την πολιτική μα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν μπορούμε να επιτύχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον ε, τους αγρότες μας. μα. Μπορούν να αποτελέσουν μέρο του προβλήματο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι κάτι τέτοιο. Απαραίτητο όμω θα πρέπει να αποτελούν, αποτελέσουν μέρο τη λύση. Ε, για να είμαστε επιτυχεί. Ε, και ε, το είχα αναφέρει ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βασιστεί στη διασφάλιση ακριβώ του εφοδιασμού με τρόφιμα των πληθυσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα ο στόχο μα είναι για αυτή τη χιλιετία να έχουμε βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και εφοδιασμό των πολιτών μα με τροφίμα. Και ακριβώ, η πρωτοβουλία από το αγρότημα στο ε, πιάτο εξετάζει αυτές τις πτυχές. Ε, σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε λιπάσματα και φυτοφάρμακα, πώ μπορούμε να μειώσουμε τις σχετικέ εκπομπές, σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε, ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης τους αλλού. Ε, τι συμβαίνει σε σχέση με τις ζωοτροφές και πώς αυτές επηρεάζουν ε, τους στόχους μας σε άλλου τομεί, για παράδειγμα τον στόχο της μείωσης της αποψήλωσης. Άρα λοιπόν η ασφάλεια ε, του εφαρμοσμένου των τροφίμων για τους πολίτες μας τα εγγυάται όλα αυτά. Και η πιο περιπλοκή πτωχή του ερωτήματος που θέσατε είναι το εξή. ότι κάποιο θα μπορούσε να πει δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα τροφίμων ε, με τις χαμελότερες ε, τιμές. Ε, ίσως δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε άλλου είδους τιμές, αλλά ερωτήστε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χρήματα για να ξοδέψουν περισσότερο σε ό,τι αφορά τα τρόφιμά τους. Δηλαδή, ε, ε, τα πράγματα έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή δεν εξασφαλίσουν το απαραίτητο εισόδημα για τους αγρότες μας. Ε, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξής μας εάν δεν συμμετάσχουν και οι αγρότες μας εδώ. Και εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν την υποστήριξη αλλά και ένα ε, ίσους του παιχνιδιού, δίκαιο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και για τους αγρότες μας. Και νομίζω πως αυτή η μετάβαση που ξεκίνησε με τον Φιλ Χόγκαν μας έχει βάλει σε σωστή ε, πορεία. Συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια ακολουθώντας τις αρχές που βάλει ο Φιλχόγκ. Ναι, να σας πω ότι δεν ε, γνωρίζω ακριβώς ε, το πώ θα συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία σα από το αγρόκτημα στο πιάτο με την αγροτική πολιτική, γιατί υπάρχει τεράστια αλληλεπικάλυψη και δεν απαντήσατε πλήρω στο ερώτημα που έθεσα. Ε, έχω δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Γιατί ε, επί της αρχής έχετε δίκιο ότι δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλά τα εισοδήματα των αγροτών. Κάποιοι βγάζουν πολλά, αλλά οι περισσότεροι βγάζουν πολύ λίγα. Ε, και όλοι μας, ε, όπως είπατε στα εισαγωγικά σας σχόλια, θα θέλαμε να επιστρέψουμε στην Επέτρο, αλλά χρειαζόμαστε και ένα εισόδημα για να το κάνουμε. και τι λέτε λοιπόν ε, ως κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνο και για το μέλλον τους οικονομικά γιατί ε, τους είπαμε για παράδειγμα να σταματήσουν να ε, τη χρήση των λοιπασμάτων τους ε, και να, κάνουν, να, μεταβάλουμε αντίστοιχο τρόπο της καλλιέργησης τους. Ε. Τώρα λοιπόν πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του αγρότε μα για να κάνουν αυτή τη μετάβαση που του ζητάτε. Απάντηση. Ναι, εγώ νιώθω τη δέσμευση να συζητήσω, να ακούσω του αγρότε μα και να του παρουσιάσω αυτή την πρωτοβουλία από το αγρότη μα στο πιάτο για να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε τα λοιπάσματά μα, πώ μπορούμε να μειώσουμε τι εκπομπέ μα και ε, Σουκομανσχολ χρειάστηκε ε, να κάνει το ίδιο, δηλαδή να ε, πείσει τους αγρότες και αυτό έγινε και στη συνέχεια. Δηλαδή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ξανά και ξανά χρειάζονται να γίνονται αυτές οι προσπάθειες. εγώ είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής και κατοχυρώνονται στις συνθήκες είναι ε, ισχύουν όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή θα πρέπει τα τρόφιμα που φτάνουν στα πιάτα μας να είναι βιώσιμα και ταυτόχρονα να επιτρέπουν στους αγρότες μας να παραμένουν στις ε, αγροτικές περιοχές ε, και να, έχουν, να υπάρχει μια επικοδομητική σχέση ανάμεσα στις υπαίθριες περιοχές αφενός και στις μητροπολιτικές αστικές περιοχές αφετέρου. Και δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό χωρίς να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας. Ε, σε ό,τι αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα ακριβώς αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε ότι η, η, η τιμές για αυτά τα τρόφιμα που παράγουν δεν είναι ανταγωνιστικές ε, σε σύγκριση με τα τρόφιμα τα οποία ε, εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και θα πρέπει να ε, συνομιλήσουμε με τους διεθνούς μας εταίρους εάν τα εν λόγω τρόφιμα, τα οποία για παράδειγμα εισάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν προϊόν αποψήλωσης. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και στο μέλλον, όπως το κάναμε άλλωστε και στο παρελθόν, για παράδειγμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία με την Μερκοσούρ. Ναι. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο των δύο και ενός λεπτών αντιστοίχως. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Χάβη Λόπεθ. Καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο. Και πάλι, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, εσείς ε, σήμερα επανειλημμένως αναφερθήκατε στην ανάγκη να γίνει μια δίκαιη οικολογική μετάβαση που να μην αφήνει κανέναν πίσω του. Και εμείς ως σοσιαλιστές ε, το υπερασπιζόμαστε αυτό τα τελευταία χρόνια και όχι την ανάγκη μόνο να είμαστε φιλόδοξοι για την ε, ε, ε διακοπή της χρήσης άνθρακα, αλλά και αυτή την ε, αλλαγή για τον τρόπο ζωή μας, ναι, στον τρόμο ζωή μας και αυτή η μετάβαση να είναι δίκαιη, να είναι δίκαιη που να κάνει καταμερισμό του κόστος, γιατί υπάρχει κόστος, αλλά να επιμερίζεται σωστά και τα ωφέλη που έχει θέσει εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν και ωφέλη. Και επομένω ε, θα θέλαμε λοιπόν αυτή τη δίκαιη μετάβαση. Και λέτε και για ένα ταμείο που. Θα ήθελα να ρωτήσω για το ταμείο και τα χαρακτηριστικά. Καταρχά θα θέλουμε να. Ε, εξασφαλίσουμε και κοινωνική διάσταση, όχι οι τεχνολογίες μόνο και τα υπόλοιπα. Επίσης, θέλουμε να είναι νέα κονδύλια, να μην ανακυκλώσουμε κονδύλια κοινωνικά ή περιφερειακά για το ε, Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Και τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα θέσουμε υπό όρους αυτή την ενίσχυση και αυτή τη χρηματοδότηση τη συμπλήρωση των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα. Εγώ ε, βρίσκομαι στην ευτυχή θέση ε, να το έχει απαντήσει αυτό ο Ντομπρόφσκι σήμερα το πρωί. Επομένως θα ακούσετε ότι η μέλους Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά με μία φωνή και επ' αυτού. Σίγουρα θα είναι νέα τα κονδύλια, φρέσκο χρήμα και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό, έτσι θα το αποκαλέσω, ώστε όλα τα μέσα και τα κονδύλια που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και εγώ γνωρίζω ότι, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, Κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη μετάβαση θα γίνουν για επενδύσεις ε, και για πράγματα που είναι πάρα πολύ κοντά στι αγοράς, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Juncker και το InvestEU. Επίσης θα μπορέσουμε έτσι να κινητοποιήσουμε και ιδιωτικά κονδύλια. Σε κάποιου όμως τομείς, ε, αν για παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανήλικου για να κάνουν μια δουλειά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα χρειαστεί χρόνος και δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά ε, ιδιωτικά κονδύλια για να επενδύσουν σε τέτοια πράγματα. Και επομένω θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκά κονδύλια και συγχρηματοδότηση για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ε, ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση βρέσκο χρήμα αλλά και συγχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και επίση συνδυασμό με τα διάφορα ταμεία που έχουμε, γεωργικό ταμείο, διαρθρωτικά ταμεία, ταμείο συνοχή, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μέσω τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ήταν ιδιαίτερα επιτυχία στο InvestEU να υπάρχει τεράστια πρόσβεση σε κονδύλια ώστε η μετάβαση αυτή στην πράσινη οικονομία να υλοποιηθεί. Και νομίζω ότι αυτό το μείγμα θα μα βοηθήσει να επιτύχουμε διότι όπω είπα και στην εισαγωγή μου δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό αν δεν πείσουμε τους ανθρώπους που θα πρέπει να αλλάξουν ότι αυτή η αλλαγή δεν αποτελεί απώλεια αλλά κέρδος. Πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι η αλλαγή σημαίνει απώλεια και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αντιλαμβάνονται και ότι μπορεί να έχει κέρδη όχι μόνο για καλύτερο περιβάλλον αλλά και για μια καλύτερη θέση εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, διευκρινίσατε πολλά πράγματα για τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και θα ήθελα να μιλήσω και για ένα άλλο νέο ε, στοιχείο το οποίο συζητιέται πολύ, ο μηχανισμός προσαρμογής συνόρων που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μας θα ανταγωνίζονται με θεμητό τρόπο, αλλά ε, θα αποφεύγουμε και το οικολογικό ντάμπινγκ. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της ιδέας, αλλά το θέμα είναι αν κάτι σύνθετο όπως είναι αυτό, ε, καταρχάς θα το αποδεσμεύσετε εσείς ως Αντιπρόεδρος ε, και μέσω του European Green Deal και ταυτόχρονα αν αυτό θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ε, πόσο θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύνθετο μέσο και επίσης ε, το Κοινοβούλιο ήδη είπε ότι συμφωνεί ότι κάτι τέτοιο ε, μηχανισμός προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα θα είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προπολογισμό. Συμφωνείτε επ' αυτού. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Η ιδέα μου είναι να πούμε στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς κάνουμε αυτή τη μετάβαση σε μια ήπειρο η οποία θα είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Για να γίνει αυτό θα λάβουμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο φυσικά και στην οικονομία μας. Εάν λάβετε κι εσεί τα ίδια μέτρα ή συγκρίσιμα μέτρα προ την ίδια κατεύθυνση, ωραία, θα το κάνουμε όλοι μαζί. Εάν όμω δεν κάνετε κάτι τέτοιο, τότε προφανώ δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προστατεύσουμε τη δική μα πλευρά και τη δική μα την οικονομία και επομένω θα εφαρμόσουμε ε, φόρο ε, άνθρακα στα σύνορα. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι συμβατό και με τον ΠΟΕ, θα πρέπει να το αναλύσουμε όμω. Πιστεύω ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Φανταστείτε ε, να έχουμε τη βιομηχανία του χάλιβα να παράγει χάλαβα με τη χρήση υδρογόνου. Δεν είναι αδύνατο πλέον, είναι δυνατόν. Αλλά ο χάλιβας αυτός όσον αφορά το κλιματικό κόστος θα είναι πολύ πιο δαπανηρός από τον χάλιβα ο οποίος παράγεται με άνθρακα στην Κίνα. Και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα ενό τόνου χάλιβα. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την ανισότητα. Γι' αυτό και μπορεί να χρειαστεί ένας φόρος ε, άνθρακα στα σύνορα. Για τους πρασίνους η Μαρή Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μας μιλείτε για τη δίκαιη μετάβαση, αλλά εμείς θα θέλαμε πράξεις. Η χώρα σας καταδικάστηκε για κλιματική δράση. Η Γαλλία και η Γερμανία ε, διώκονται συνεχώς από τους πολίτες και από πολλές άλλες χώρες στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου γιατί η κλιματική δράση ε, είναι και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θεωρείται. Δεν ακούω όμω ούτε φιλοδοξίε ούτε συνέχεια για αυτό το Green Deal. Πού είναι η συνέπεια όταν βάσει όλων των επιστημονικών ενδείξεων η Ευρώπη για την ε, ε, μετάβαση αυτή ε, βασίζεται σε πολλέ δυνατότητε ορικτών καυσίμων. Πού γίνεται, πού βρίσκεται η συνογή για την αποψήλωση. Χωρί, όταν εμεί εμπορευόμαστε εδώ στην Ευρώπη και στην εσωτερική αγορά τέτοια πράγματα. Πότε σκοπεύετε λοιπόν να δώσετε ένα τέλος στις άμεσες και έμεσες ενισχύσεις ε, στο φυσικό αέριο. Σκοπεύετε να προτείνετε δεσμευτική νομοθεσία για να προστατεύσετε τα δάση του κόσμου, τις περιβαλλοντικές βιαιότητες που διαπράττουν οι επιχειρήσεις μας. Όπως ε, είπα ήδη, θεωρώ ότι ένα από τα πιο ε, σύνθετα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί είναι να υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές μας. Και δεν σας κρυβώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς η ε, ίδια μου είπατε πόσο σύνθετα είναι τα θέματα αυτά. Δεν έχω καμία ψευδέστηση ότι θα υπάρξει συνέπεια μέσα σε 100 μέρες. Αλλά το να βρούμε πού βρίσκονται οι ασυνέπειες και στη συνέχεια να υποδείξουμε την νομοθεσία και τα βήματα που θα λάβουμε και όλα τα υπόλοιπα που θα κάνουμε για να ε, σταματήσουν αυτές οι ασυνέπειες θα είναι ένα από τα πιο σύνθετα καθήκοντα αλλά ένα και από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του χαρτοφυλακίου μου. Όπως ε, λέτε κι εσείς, ε, το φυσικό αέριο αποτελεί πρόβλημα. Ναι, δεν είναι βιώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά το φυσικό αέριο θα είναι τμήμα της μετάβασης που ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνουμε προς την βιώσιμη ενέργεια. Και αναφερόμαστε και στις υποδομές. Ε, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια έργα, αναφερθήκατε και στη χώρα μου, υπάρχουν έργα για να μπορέσουμε να έχουμε και μεταφορά υδρογόνου και να έχουμε κατάλληλε υποδομέ, τι οποίε μπορούμε να κατασκευάσουμε πολύ εύκολα. Και ελπίζω λοιπόν σε ένα εγγύ μέλλον να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε υποδομές οι οποίες δημιουργήθηκαν για το φυσικό αέριο για τη μεταφορά μιας μορφής ενέργειας που είναι απόλυτα βιώσιμη, του υδρογόνου. Δεν ε, πρόκειται λοιπόν μόνο για ανακοίνωση άσχημων ειδήσεων, αλλά έχετε δίκιο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ γρήγορα να ε, μην εξαρτώμαστε από την ορυκτή ενέργεια. Δεν σας κρύβω ότι θα είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω στην πολιτική και αν έχω τη δυνατότητα να αποδείξω και να βρω πού βρίσκονται οι ασυνέπειες, είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες θα υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τις επιτρέψουν ε, να διαγράψει αυτές τις συνέπειες. Έχετε απόλυτο δίκιο όμως ότι όντω υπάρχουν ασυνέπειες στι πολιτικές μας σήμερα. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Νομίζω όμως ότι θα επαναλάβω την ερώτησή μου. Θεωρείτε και αν ναι ότι πρέπει να βάλετε ένα τέλος σε αυτές τις άμεσες και έμεσες ενισχύσεις στα ορυκτά καύσιμα. Πιστεύετε ότι για τα δάση όπως και για το κλίμα θα πρέπει να δεσμεύσουμε τις επιχειρήσεις μας να δράσουμε. Για παράδειγμα για την υποχρέωση επαγρύπνεσης. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Να τους υποχρεώσουν να μειώσουν τις εκπομπές τους. Να τιμωρήσετε αυτούς που δεν τις μειώνουν. Και επίσης να απογορεύσετε και να τιμωρήσετε ώστε να προλάβουμε και... Ε, περιβαλλοντικά εγκλήματα και οικοεγκλήματα. Ευχαριστώ που θα απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Αυτά όλα, είναι όλα. Ναι, σκοπεύω να λάβω τα μέτρα για τις ενισχύσεις για την ενέργεια, ε, τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας, ε, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση να σας δώσω σήμερα. Θα δώσω αυτές τις απαντήσεις όταν θα αναλύσω και τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες που έχουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μάλλον περιορισμένες, αλλά εμείς θα την κάνουμε την ανάλυση αυτή. Ε, καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σας, είναι λογικό, είναι συνεκτικό, αλλά δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση να σας δώσω. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που ρωτάτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να ε, προστατεύσουν προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, και το πώς ε, ε, επηρεάζουν οι δράσεις τους στην βιοπικιλότητα, πιστεύω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την απαραίτητη διαφάνεια για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, ώστε να γνωρίζουν αν ένα προϊόν δημιουργήθηκε ει βάρο των δασών, ει βάρο τη βιοπικιλότητα ε, και μέσω αποψήλωση. Είναι ένα πρώτο βήμα, μπορεί αυτό να γίνει με την επισήμανση, μπορεί να γίνει και με άλλα μέτρα, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και απαγόρευση, αλλά προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει μια πιο ει ανάλυση του αντικτύπου και ε, αν μπορώ να προτείνω κάποια μέτρα για τα πλαστικά ή για τα απόβλητα και μπόρεσα να το κάνω την προηγούμενη πενταετία ήταν γιατί έγινε μια ανάλυση των συνεπειών πρώτα και μπόρεσα να προτείνω κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ήταν συνεπές. Δεν θέλω να προχωρήσω λοιπόν πολύ βιαστικά και να σας κάνω συγκεκριμένες προτάσεις τώρα. Θα γίνω την ανάλυση, αλλά κατάλαβα απόλυτα τι λέτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να λάβει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από μια ανάλυση που θα μας ε, δείξει ποιος είναι ο αντίκτυπος. Η κυρία Ωρέλια ID. Κύριε η κυρία Φοντερ Λάιεν μας παρουσίασε μια στρατηγική για τη βιοπικιλότητα για το 2030. Μεταξύ των στόχων λοιπόν που έχει, αν θα θέλετε να πλησιάσετε το μικρόφωνο, λέει ο Πρόεδρος, να ξαναξεκινήσω λοιπόν. Η κυρία Φοντερ Λάιεν μας παρουσίασε λοιπόν μια στρατηγική για τη βιοπικιλότητα για το 2030 και ανάμεσα στους στόχους που παρουσιάζει θέλει να βάλει τέρμα στην απώλεια βιοπικιλότητα σε ό,τι αφορά την καταστροφή βιοσυστημάτων Παραδόξως όμως, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ανανεώσιμες ε, ενέργειες ε, ε, μα οδήγησε στην αποψήλωση των τροπικών δασών. Και να μην ξεχνάμε κυρίως τις ελεύθερες και εμπορικές σχέσεις σε ό,τι αφορά αρνητικές συνέπειες των περιβάλλων. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για να κινηθούμε προς μια οικονομία βιώσιμη και με ποιους όρους σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, έλαβα σήμερα το απόγευμα, Από οι δικέ σα, σε ό,τι αφορά την έλλειψη συνοχή που υπάρχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Γιατί έχουμε εισαγάγει πολιτικές σε πολλέ περιπτώσει ε, με καλές προθέσεις, με αποτέλεσμα όμω αντίθετο από το αποσκοπούμενο σε κάποιους άλλους τομείς. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για μένα αυτό που θα είναι σημαντικό και θα είναι μεγάλο τμήμα της δουλειά μου, είναι να εξασφαλίσω συνοχή στις πολιτικές. Δεν βλέπω ωστόσο να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των όσων ε, λέτε για τη βιοπικιλότητα και την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω ότι τα δύο αυτά στοιχεία λειτουργούν ε, συμπληρωματικά. Πείτε μου λοιπόν, πού θεωρείτε ότι υπάρχει αντίφαση. Αν ε, μου δείξετε κάτι τέτοιο, θα είμαι στη διάθεσή σας να δω πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η μείωση των εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου και η μείωση της ε, αύξηση του κλίμα, της θερμοκρασίας, η μείωση της απώλειας της βιοπικιλότητας είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί από κοινού και μάλιστα κατεπηγόντως. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη αυτή ανάπτυξη, σε ποιο χρόνο διάγραμμα θα κινηθείτε σε ό,τι αφορά τα ορεικτά καύσιμα, την κατάργηση αυτών και την κατάργηση των επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία αυτή. Σε ό,τι αφορά την ε, μείωση της, ε, του άνθρακα που επιθυμεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν θα δημιουργήσουμε αρνητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει μα και θα ενθαρρύνουμε τι εισαγωγέ. Απάντηση. Είναι πραγματικά αναπόφευκτο και απαραίτητο να μειώσουμε τις επιδοτήσεις και να τις κατηγορήσουμε τις επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Θα πρέπει να καταρτήσουμε συγκεκριμένο σχέδιο για συγκεκριμένα βήματα, τα οποία θα κληθούμε να τα συζητήσουμε με τα κρατημέλη. Αλλά υπάρχουν ε, προφανείς ε, αντιφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις απαλείψουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το διεθνές εμπόριο που αναφέρεται στη διάσκεψη στην Κίνα για την βιοπικιλότητα, αλλά και στις διαπραγματεύσεις τις οποίες θα κάνουμε για τις εμπορικές συμφωνίες, με το Μερκοσούρ, για παράδειγμα. Υπάρχει επιθυμία να υπάρξουν ε, εισαγωγές προ την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε να κινηθούμε. Αυτό είναι επισημία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το Μερκοσούρ, για παράδειγμα, ε, υπάρχουν ε, περιορισμοί για τη Βραζιλία, για παράδειγμα, για να πετύχει του στόχου και να τηρήσει του στόχου του Παρισιού. Και αυτά θεωρώ ότι είναι επιτεύγματα για το κλίμα και μάλιστα πολύ σημαντικά. Σα ευχαριστώ για το ECR τώρα, η κυρία Ζαλεύσκα. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω Κύριε Τιμέρμαν, θα ήθελα να θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, γνωρίζουμε συχνά ότι καλές προθέσεις ε, τελικά μπορεί να μην οδηγήσουν πουθενά. Ε, προσδοκίες των νέων μας ε, είναι πολύ υψηλέ. Ε, Θέλω να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και να αναφερθείτε και στις συγκεκριμένες χρηματοδοτικές πηγές για όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, πρώτο συγκεκριμένο ερώτημα που ε, θέλω να σας θέσω σε ό,τι αφορά ε, το νέο νόμο για το κλίμα, τον οποίο θέλετε να προτείνετε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Πώ ακριβώ θα είναι διαμορφωμένος, τι θα περιλαμβάνει και πώς θα υποβοηθήσει αυτόν τον στόχο του 40% ο οποίος ακόμα δεν έχει επιτευχθεί από μια σειρά από κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, δηλαδή, πώς θα σχετίζονται οι στόχοι αυτού του νέου ε, νόμου για το κλίμα με τους ε, παλαιότερους ε, στόχους και στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της λογικής του one in, one out που αναφέρθηκε. Τι δηλαδή θα αφαιρεθεί αν θέλετε από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ισχύσει ο νέος ε, ε, νόμος. Μετά ε, αναφέρεστε στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης αλλά έχουμε μόνο 5 δισεκατομμύρια προβλέψει για όλους τους τομείς. τι μπορούμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά. χρειάζεται δηλαδή μόνο και μόνο η Πολωνία εκατοντάδες εκατομμυρίων σλότη μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιτύχει αυτή τη μετάβαση. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσετε και... Συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βέβαια καλείται να υποστηρίξει φιλοπεριβαλλοντικά ε, project, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει και έργα για το φυσικό αέριο. Απάντηση. Ε, ο νόμος για το κλίμα θα θέσει δεσμευτικά τον στόχο του να έχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2050 και από εκεί και μετά θα δούμε ποιοι είναι διάμεσοι στόχοι τους οποίους θα επιτύχουμε για να φτάσουμε εκεί. Άρα λοιπόν ο νόμος για το κλίμα θα μας δώσει τη σαφήνεια ως προς το ποια θα είναι τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το νομικά πλέον δεσμευτικά στόχο. Ε, τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη λοιπόν στο πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων δράσης. Και νομίζω πως ε, αυτό θα αποτελέσει και αναπόσπαστο στοιχείο του ενεργειακού μείγματος για τις επόμενες δεκαετίες, πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ πως ε, και στην Πολωνία υπάρχει μαζική υποστήριξη από την πλευρά των πολιτών να αναλυφθεί δράση σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θα πρέπει να αναλυφθεί η δράση και πραγματικά με ενθαρρύνουν πολύ και όλες οι έρευνες οι οποίες διεξάγονται στην Πολωνία και με ενθαρρύνουν και οι νέοι και η στάση τους ε, στην Πολωνία. Το είπατε κι εσείς ότι πραγματικά δραστηριοποιούνται ε, και το θαυμάζω πολύ αυτό. Και ε, πραγματικά πιστεύω ότι ο νόμος για το κλίμα θα μας παράσχει το απαραίτητο πλαίσιο έτσι ώστε να πειθαρχήσουν τα κράτη-μέλη και να καταρτήσουν πολύ συγκεκριμένα σχέδια δράσης, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τα διαφορετικά στάδια τα οποία θα πρέπει να διατρέξουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στο στόχο του 2050. Υπάρχουν, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ανταποκριθεί στους στόχους μέχρι τώρα, αλλά κάποια όλα, αλλά όχι, οπότε θα πρέπει να θέσουμε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του one in, one out, ε, Μαρκος Σεύκοβιτς ήδη αναφέρθηκε, ενδεχομένω όχι ενώπιον σα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια γενική προσέγγιση, την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και το ανέφερα και εγώ πριν από πέντε χρόνια, ότι δηλαδή ε, δεν έχουμε να κάνουμε με απορρίθμιση εδώ με χαμηλότερα πρότυπα, θέλουμε καλύτερη νομοθεσία. Δηλαδή θέλουμε ψηλότερα πρότυπα, όχι χαμηλότερα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερη επιβάρυνση, λιγότερο διοικητικό άκτο για όσους ε, έχουν να κάνουν με, αυτές τις, με αυτά τα κανονιστικά πλαίσια, με αυτούς τους ε, νόμους. Και Πράγματι έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα στο πλαίσιο και της ε, ε, συμφωνίας για την καλύτερη νομοπαραγωγή, αλλά νομίζω πως μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Σε κάθε όμως περίπτωση, ναι, θα χρειαστεί νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα το αναλάβει από μόλι τη αγορά. Ναι, θα χρειαστεί νομοθεσία και μάλιστα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δευτερολογία, κυρία Ζαλεύσκα. Ναι, ε, κύριε Τίμερμαν, δυστυχώς δεν μου δώσατε συγκεκριμένες απαντήσεις. Δηλαδή δεν δίνετε απαντήσεις σε ό,τι αφορά ε, τις χρηματοδοτικές επιτυχίες. Ε, και συγκεκριμένα και για το νόμο για το κλίμα δεν μου απαντήσατε το συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσα. Γιατί ε, εδώ προσπάθησα να σας εξηγήσω λίγο τις αντιφάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, το πακέτο για την κινητικότητα συμφωνήθηκε, μετά από πολύ μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ καν στο πώς έτρεξαν αυτές οι διαπραγματεύσεις γιατί δεν είχαν να κάνουν τίποτα με μια δίκη ε, νομοθετική διαδικασία αλλά τελικά το αποτέλεσμα αυτού του πακέτου ε, θα είναι υψηλότερε εκπομπές γιατί ε, τα μεγάλα φορτηγά θα πρέπει ε, τελικά να επιστρέφουν χωρίς ε, ε, στις, ε, στα σημεία από τα οποία ε, προέρχονται, πράγμα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί επιβάρυνση. Ο κύριος Τιμερμάν, απαντά, υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο, ζητώ συγγνώμη προσπαθούσα να σας βρω, έχουμε λοιπόν το συγκεκριμένο κονδύλι το οποίο έχουμε προβλέψει και είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι για την δίκαιη μετάβαση ειδικότερα στις χώρες εκείνες οι οποίες εξαρτώνται πολύ από τον τομέα του άνθρακα, θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα κονδύλια από αυτά του ε, Ταμείου για την ε, δίκαιη μετάβαση. Αλλά θα πρέπει να είναι και ξεκάθαρο το γεγονό ότι δεν υπάρχει πλέον μέλλον σε αυτό το τομέα του άνθρακα, οπότε θα πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή οι περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από αυτό το κλάδο, είτε είναι στην Πολωνία, είτε στη Σλοβακία, είτε είναι στην Ισπανία, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, θα πρέπει να επωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη γιατί θα πρέπει να κάνουν αυτή τη μετάβαση όλες αυτές τις περιοχές θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και να εξετάσουμε ε, και τα εφιστάμενα ταμεία έτσι ώστε να ε, υπάρξουν και στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση της δίκαιης μετάβασης ε, που θα επιτευχθούν. δεν επιτύχαμε δηλαδή πολλά πράγματα στο πλαίσιο των διαφορετικών ταμείων και στην Πολωνία δεν είδατε δηλαδή πόσο έχει μετασχηματιστεί η κοινωνία στην Πολωνία και του ρυθμού ανάπτυξη, του οποίου ζηλεύουν πολλά άλλα κράτη-μέλη, του οποίου επιτυγχάνει σήμερα η Πολωνία. Α ε, κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για την ε, Πολωνία. Είναι υποχρεωμένη και θα είναι επώδυνη αυτή η διαδικασία τη μετάβαση και τη εξόδου από το άνθρακα για την Πολωνία. Αλλά εμεί θα κάνουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να το κάνει με το λιγότερο επώδυνο τρόπο και σας το λέω αυτό δηλαδή πραγματικά ως ε, εγγονός ανθρακορίχων. Κυρία από το ΕΛΚΑ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμη κυρία Τίμερμαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει ισχυρή βιομηχανική βάση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίε στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη ευτυχώς συνεχίζουμε να φτιάχνουμε ε, αυτοκίνητα, χαρτί, χάλιβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα, πολλά ακόμα. Αυτό ξέρω το Θεό. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν με την ε, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να μην μεταφερθεί ένα τμήμα τη βιομηχανή τη Ευρώπη εκτό Ευρώπη. Πώ θέλετε λοιπόν να πετύχετε η ευρωπαϊκή βιομηχανική μα βάση, οι επιχειρήσει μα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει που α, θα πληχθούν από την Πράσινη Συμφωνία τελικά να μην αποδυναμωθούν, να ενισχυθούν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω γιατί αναφερθήκατε στον φόρο για τον άνθρακα στις γραπτές σας απαντήσει. Δεν νομίζω ότι θα αποτρέψει αυτό την ε, εγκατάλειψη των επιχειρήσεων της Ευρώπης από τις επιχειρήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι πριν από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη είχαμε 5 μεγάλους παραγωγούς ε, στην Ευρώπη. Ε, πλέον δεν υπάρχει καμία μεγάλη τέτοια επιχείρηση στην Ευρώπη. Και αυτό προφανώ έχει συνεπεί και για τι θέσει απασχόληση. Όταν μιλώ με εκπροσώπου του κλάδου, απάντηση. Όλοι συμφωνούν ότι αυτή η μετάβαση είναι απαραίτητη. Και νομίζω ότι η Ήπειρο ε, που θα κάνει πρώτα τη μετάβαση αυτή θα είναι αυτή που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι όσο πιο πολύ επιμείνουμε και στηριχθούμε σε αυτή την παλιά βιομηχανία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι η μετάβαση. Εμείς στην Ευρώπη λοιπόν θεωρώ ότι είμαστε οι πιο ανταδειγμένοι να οργανώσουμε τα πράγματα σε ένα επίπεδο το οποίο θα έχει νόημα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την βιομηχανία μα, αλλά στι πιο πολλέ περιπτώσει θα πρέπει να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την βιομηχανία μα, προκειμένου να απελευθερωθεί από τα δεσμά τη εξάρτηση από τι ε, παλιέ ε, πηγέ ενέργεια. Αυτό το ανέφερα ότι ακόμα και η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλιβα κάνει έντονες προσπάθεια να επεξαρτοποιηθεί, να από τις ατορικά κόψιμα, για παράδειγμα, των υδρογόνων. Πώς μπορούμε με υδρογόνο να κάνουμε να φτιάξουμε χάλιβα. Αυτό πριν από 5-6 χρόνια ήταν αδιανόητο και τώρα είναι σχεδόν ρεαλιστικό. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει κατανοήσει ότι αυτή η μετάβαση είναι απαραίτητη και για τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Το διαπιστώνουμε ήδη στι ΗΠΑ όχι σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά οι επιχειρήσεις, οι πολιτείες είναι εκείνες που έχουν κατάληξει στο ίδιο συμπέρασμα. Και στην Κίνα το βλέπουμε αυτό, όπου τα πράγματα αλλάζουν δραστικά και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Και εμείς έχουμε χάσει την ευκαιρία αυτή. Έχουμε χάσει την ευκαιρία του διαδικτύου, του ίντερνετ. Λέγαμε ότι το θέμα ήταν οι τηλεπικοινωνίες και όχι το ίντερνετ. Και αυτό ήταν τεράστιο σφάλμα. Αυτό που δεν έχουμε χάσει όμως είναι η ευκαιρία της βιώσιμης βιομηχανίας και πιστεύω ότι εδώ η Ευρώπη έχει πολύ καλές ευκαιρίες και δυνατότητε να προχωρήσει εδώ και να αναξερτοποιηθεί από τις dark καύσιμα αν φροντίσουμε, αν φροντίσουμε όλα αυτά που αφευρίσκουμε τώρα να μπορέσουν να προσανατολιστούν στο 5G. Η αυτοκίνητο βιομηχανία μας να αναξερτοποιηθεί από τους κλασικούς κινητήρες, να φροντίσουμε οι υποδομές μας να βελτιωθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά τους συντεροδρόμους. Έχουμε τεράστια καθήκοντα και πολύ μεγάλα πράγματα να κάνουμε. Αυτό είναι καλό για τη βιομηχανία. Είμαι αισιόδοξο, ξέρετε, ότι μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Γιατί είμαι και απόλυτα πεπισμένο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ απλό. Όποιος το πετύχει αυτό πιο γρήγορα θα έχει τις καλύτερες ε, ευκαιρίες. Και αυτό προκύπτει από όλες τις μελέτες, ότι θα πετύχουμε επιπλέον ανάπτυξη στην Ευρώπη αν κάνουμε γρήγορα τη μεταβάση αυτή. Η κυρία Νίμπλερ. Ε, καλή αισιοδοξία σας και ελπίζω να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Κάναμε τη συζήτηση εδώ και ακούσαμε πολλά για πολλοί κανονισμούς και ρύθμιση. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό αυτό. Να υπάρχουν χρήματα για την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν το άκουσα αυτό καθόλου. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Το αναφέρατε σε ό,τι αφορά το 9% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων που προκύπτει από την Ευρώπη σήμερα. Και η ΕΠΑ που είναι ο πιο μεγάλος ε, υπεύθυνο για τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου έχει φύγει και έχει καταλήξει την συνθήκη των Παρισίων και η Κίνα ε, εξαρτάται από το δολάριο για την οικοδόμηση τέτοιων εργοστασίων ε, ανθρακά. Τι κάνετε λοιπόν εσείς προκειμένου σε παγκόσμιο επίπεδο να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί οι μεγάλοι φορείς εκπομπών. Ε? Όπως σας είπα, απάντηση. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι ενδεχομένως να πετύχουμε συμφωνία με τους Κινέζους. Προς την κατεύθυνση αυτή θέλουν να κινηθούν. Σε ό,τι αφορά τις είπα τώρα, θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του ομοσπονδιακού επίπεδου και των δηλώσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο και των ε, συμφωνιών με τις πολιτείες και με τις μεμονωμένες πόλεις. Εδώ υπάρχουν πολλοί σύμμαχοι που γνωρίζουν πολύ καλά προς τα που πρέπει να οδεύσουμε. Αλλά να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι και εγώ ε, αισθάνθηκα πριν από κάποιες εβδομάδες όταν μετέβησα στην Νέα Υόρκη ότι τα, οι μεγάλες βιομηχανικές πολιτείες δεν κινητοποιούνται ε, επαρκώς σε ό,τι αφορά ε, την πράσινη μετάβαση. Έχουμε λοιπόν τεράστια δουλειά να κάνουμε σε ό,τι αφορά το να πείσουμε και τους υπόλοιπους. Ε. Επαναλαμβάνω όμως ότι πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να γίνει. Αν καθυστερήσουμε όμως, δεν θα το πετύχουμε αυτό. Δεν θα το καταφέρουμε. Υπάρχουν κάποια σημεία καμπής, λοιπόν. Δεν θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό. Νομίζω λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια έχουμε τεράστιο έργο και θα πρέπει να πείσουμε τους διεθνείς μας ατέρους. Με την Κίνα είμαι μάλλον αισιόδοξο και νομίζω ότι και στις είπα κάτι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά πραγματικά είναι γιγάντιο το έργο. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Okay, Κύριε Τίμερμαν, σας παρακαλώ να κρατάτε το χρονομιλία σας. Ο Γιάννου Ήτεμα τώρα από το Ρενιού, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ κάθομαι, κύριε Τίμερμαν. Μιλήσαμε για την ε, κανονισμούς, για το προπολογισμό και τώρα, όπω είπε και η προηγούμενη ομιλητρία, δεν ακούσαμε τίποτα για την καινοτομία, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν νέε ιδέε, οι οποίε δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για του στόχου, για το κλίμα και για το περιβάλλον. Αυτό συχνά όμω που βλέπω είναι ότι υπάρχουν παροχημένε νομοθεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 30 χρόνων και παραπάνω, που ε, είναι αντιφατικέ με του στόχου μα. Και αυτό που χρειάζεται είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πειραματιστούμε σε ό,τι αφορά τις νέες αυτές ιδέες, τις καινοτομίες. ερωτώ λοιπόν, πώς θα προωθήσετε αυτό το κλίμα και αυτή την ατμόσφαιρα καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις νέες φύσεις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ταμπού σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα, ή την βιοτεχνολογία. Απάντηση. Δεν έχουμε κανένα ταμπού. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη όλα αυτά να τεκμηριωθούν με επιστημονικό τρόπο και μάλιστα απόλυτα. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια γίνονται πολλές επενδύσεις και σε θέματα ασφάλειας και όπως ξέρετε υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε όμως όταν μιλάτε για την αντίφαση μεταξύ νομοθεσίας και καινοτομίας Πιστεύετε πραγματικά ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία θα υπήρχαν οι καινοτομίε που υπάρχουν ε, τα τελευταία χρόνια, αν δεν είχαν αντιμετωπίσει τι τεράστιε περιορισμού σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ, νομίζω ότι δώσαμε τεράστια όθεση στην καινοτομία. Αντιθέτω, και επιταχύναμε κάτι το οποίο έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους κανονισμούς, θεωρώ ότι μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν την καινοτομία του τουλεχθέντος. Πιστεύω ότι όπως και στο παρελθόν θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο περιθώριο και μεγάλο ε, περιθώριο ανάπτυξη στην καινοτομία. Και αυτό λειτουργήσε πολύ καλά και στην Ολλανδία, από ό,τι ξέρετε. Και ξέρουμε ότι ε, και στον τομέα αυτό συγκαταλέγονται και πολλά έργα ανανεώσιμων ενεργειών, πηγών ενεργειές. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Όλα αυτά τα έργα λοιπόν που προέκυψαν Πρόσφατα άκουσα και για μία καινοτομία όπου με ηλιακά πάνελ μπορούμε να ζεστάνουμε νερό χωρίς ε, ηλεκτρισμό. Φανταστείτε ότι μιλάμε για τέτοια έργα μικρής κλίμακας τα οποία στη συνέχεια αναβαθμίζονται. Είναι εντυπωσιακό. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσουμε και το θέμα των ε, νεοφιών επιχειρήσεων. Να υπάρχουν αυτές οι επαφές γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τον επόμενο καιρό. Και εδώ είναι η δύναμη της Ευρώπης. Η ανανεώσιμη πηγή της ενέργειας δεν μπορεί να μεταφερθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τοπικό επίπεδο, στην στέγη, στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι. Και αυτό έχει άμεσα αποτελέσματα και άμεσα θετικέ συνέπειες για τις θέσει απασχόλησης, κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει στην Ευρώπη. Και ερώτηση. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να ξέρει ο κόσμο, για να μα εμπιστεύεται, ότι δεν επενδύουμε σε πράγματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Και θα ήθελα επίση να τονίσω ότι αυτό θα πρέπει να μπορεί να το πληρώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ε, φοβούνται πάρα πολύ ότι θα χρεοκοπήσουν. Για παράδειγμα, στη Γεωργία ε, δημοσιεύτηκε μια ε, έρευνα στην ε, Ολλανδία ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να τα βγάζουν πέρα. Πώ θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτά, γιατί πολλοί αγρότε θέλουν να πετύχουν κάτι καλύτερο, θέλουν να κινηθούν προ την ε, βιολογική γεωργία, αλλά πολύ απλά δεν υπάρχει ζήτηση από την αγορά για να καλυφθεί το έξτρα κόστο αυτό. Και όταν υπάρχει το θέμα τη μίση των τιμών α, λόγω των παγκόσμιων τιμών, απάντηση. Όπω είπα και προηγουμένω προ την κυρία Μαγκίνε στο επίπεδο αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω και πολλά δεν έχουμε κάνει. Και επειδή ο αγροτικός κλάδος ε, οι αγρότες είναι έξυπνοι, καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση και σε κάποιες περιπτώσεις όμως ε, είναι τόσο μεγάλη αυτή η μετάβαση που βγαίνουν στους δρόμους και δεν δηλώνουν, δεν καταλαβαίνουν πώς πρέπει να γίνει η μετάβαση. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και να πούμε ότι κοιτάξτε μπορούμε να κάνουμε αυτό για παράδειγμα με τα λοιπάσματα, μπορούμε να κάνουμε αυτό το χύψη σε ό,τι αφορά την κοινοτομία για τη μείωση των εκπομπών, σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, σε ό,τι αφορά τις νέες καλλιέργειες. Να δώσουμε λοιπόν κατασυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά α, τα πλεονάσματα στη γεωργία και στην υιοτροφία, που προκαλούν βλάβες και στην φύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, να τα διευκρινίσουμε πολύ περισσότερο τα τελευταία επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να δώσουμε μια προοπτική στον αγροτικό κλάδο στην Ευρώπη για να υπάρχει βιωσιμότητα και αυτό θα πρέπει να είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τους μη εγγεγραμμένους η Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ είμαι. Καλησπέρα σας. Εγώ επανέρχομαι στο επωνόδημα, ε, επωνίδη στο θέμα των ενισχύσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Το θίξατε, αλλά θα ήθελα να το θίξω και εγώ, γιατί ακόμα υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 55 δις το χρόνο πηγαίνουν ακόμα σε ενίσχυση στα ορυκτά καύσιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο μέρος της ευθύνη είναι των κρατών μελών και τα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που παρουσιάστηκαν δεν είναι αμφίσιμα, είναι, δεν είναι φιλόδοξα, συγγνώμη, είναι αμφίσιμα, ε, συγκεχημένα για το το τι σκοπεύουν να κάνουν τα κράτη-μέλη για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τέτοιε πηγέ ε, το συντομότερο δυνατόν. Ευτυχώ υπάρχουν κάποιε καλέ εξαιρέσει και η Ιταλία ε, πλέον είναι μεταξύ των χωρών που αποτελούν εξαίρεση. Έχουμε όμως ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Θα ήθελα να ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα ενώπιον των κρατών μελών επ' αυτού για να επιταχύνουμε αυτή την τόσο απαραίτητη ε, διακοπή της χρήσης αυτών των καυσίμων. Επίση, ξεκινώντα από τι μεγάλε διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, κάποια είναι σε θέση να κάνουν πολλέ επενδύσει χωρί πολλέ θυσίε, ενώ κάποια άλλα κρατημέλη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εσείς ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει όλοι να είναι σε θέση ε, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, κατεπηγόντω τι κοινωνικέ και κλιματικέ προκλήσει. Μήπως έχει φτάσει η στιγμή να αλλάξουμε τις φορολογικούς κανόνες και τους δημοσιονομικούς κανόνες και να αποκλείσουμε τις ενισχύσει αυτές ε, στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη. ώστε επιτέλους να μην ε, υποστηρίζουμε αυτές τις μορφές. Εγώ θα έλεγα ότι εάν θέλουμε να φτάσουμε όλοι, όπως λέγεται στα Ιταλικά, πώς λέγεται τώρα στα Ιταλικά η ουδετερότητα του άνθρακα, ε, Αν όντω λοιπόν θέλουμε να έχουμε κλιματική ουδετερότητα το 2050, θα πρέπει όλε οι χώρε να έχουν σχέδια για το πώ θα το πετύχουν. Αν έχουν τέτοια σχέδια, θα πρέπει να πούνε και τι θα κάνουν με τι παραδοσιακέ μορφέ ενέργεια. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τα βοηθήσουμε ε, να κάνουν επενδύσει ε, και να μην κάνουν επενδύσει προ την αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ λοιπόν ότι θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το εργαλείο για να έχουμε ένα σχέδιο με τα κράτη-μέλη για ε, να προχωρήσουμε και να ε, έχουμε κλιματική ουδετερότητα για το 2050. Για τη δεύτερη ερώτηση που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, αποκλεισμό των πράσινων επενδύσεων από τον ε, υπολογισμό του ελλείμματο για το ε, σύμφωνο σταθερότητα. σω επειδή είμαι Ολλανδό, μου διέφυγε αυτή η ερώτηση. Τέλο πάντων, πέρα από τα αστεία. Πιστεύω ότι σήμερα ο Βαλτής Δομπρόσκης ε, έδωσε κάποιες ενδείξεις επ' αυτού. Νομίζω ότι όταν εξετάζουμε την οικονομική ανάπτυξη των ε, κρατών μελών μας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλα εκείνα τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε μια βιώσιμη κοινωνία. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει τμήμα της ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, αλλά εγώ δεν προτείνω να αποκλείσουμε κάποιες επενδύσεις ε, έτσι στον αέρα από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, ευχαριστώ παρόλα αυτά για την απάντησή σας. Να περάσω σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά ένα θέμα το οποίο έχετε θίξει ήδη, την στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, διότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερε επιστημονικέ ενδείξει που μα αποδεικνύουν ότι η εντατική καλλιέργεια, κυρίω η βιομηχανική κτηνοτροφία, ε, πιέζουν και τη βιοπικιλότητα αλλά και τι εκπομπέ ε, αερίου του θερμοκηπίου. Θα φροντίσετε λοιπόν εσείς ε, να επανέλθω και πάλι στο θέμα της χρηματοδότησης, να μην χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για να χρηματοδοτούμε ε, εντατική κτηνοτροφία, αλλά ίσα ίσα να ε, ενθαρρύνουμε μικρότερη κατανάλωση ζωικών προϊόντων, αλλά καλύτερες ποιότητας και περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία κάνουν και οι ίδιοι οι γεωργοί και εκτινοτρόφοι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιβάλλουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο ζητούν αυτοί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την κοινή αγροτική πολιτική από αυτό το πρίσμα. Να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε ένα μέλλον στους Ευρωπαίους παραγωγούς βάσει ε, τροφίμων τα οποία θα είναι σωστά και δεν θα ρηπαίνουν η εντατική καλλιέργεια θα διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό είναι ήδη τμήμα των μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής Juncker, αλλά θα αποτελέσει και τμήμα της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο, ε, στο πιάτο. Τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η Σιμώνα Μποναφέ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο ναι μεν συζητήθηκε ήδη, αλλά θεωρώ ότι είναι κεντρική σημασία. Είναι η άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Green Deal και της, ε, των επενδύσεων που εφαρμόζονται. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Green Deal, θα πρέπει να δράσουμε οριζόντια. Το είπατε ήδη, σε πολλούς τομείς. Ε, σκέφτομαι τον τομέα της, ε, των μεταφορών με βιώσιμες υποδομές, ε, τη βιομηχανία επίσης, ε, παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους μας, αλλά ε, και μέτρα τα οποία αναφέρατε κι εσείς, η στήριξη των εργαζομένων που εργάζονται σε ιδιαίτερα ρηπογόνους τομείς και μέτρα για νέες δεξιότητες ώστε να αλλάξουν και να πάμε σε νέα επαγγέλματα. Αυτό απαιτεί νέες επενδύσεις και νέους πόρους και μόνο με τη Συμφωνία των Παρισιών υπολογίζεται ότι χρειαζόμαστε από 180 έως 200 δις ευρώ το χρόνο. Εσείς αναφερθήκατε στις ιδιωτικές επενδύσεις, στις επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη συγχρηματοδότησης με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά χρειάζονται και πάρα πολλοί δημόσιοι, ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Ποιε είναι οι ιδέε σα ώστε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού προπολογισμού το οποίο θα χρηματοδοτήσει πραγματικά το Green Deal. Εγώ όταν αναφέρομαι στο Ταμείο δίκαιη Μετάβασης εντό της ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρομαι και σε ένα μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι κάνουμε θα γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εδώ αναφέρομαι σε όλα τα ταμεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Και εδώ φρονώ ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά, διότι όπως γνωρίζετε τα τομεία έχουν τη δική τους λογική. Ορισμένες φορές έχουν ήδη ενσωματώσει και εντάξει το γεγονός ότι πρέπει να δίνουν 25% ό,τι κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το ιδεώδες για μένα θα ήταν να δίνεται το 100% των κονδυλίων για να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση όλοι και τουλάχιστον ως πρώτο βήμα να αποφύγουμε να κάνουμε πράγματα που πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα μπορούμε να το εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Έχετε δίκιο λοιπόν εσείς. Μόνο για την ε, Συμφωνία των Παρισιών χρειαζόμαστε 200 δις το χρόνο. Αν ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την ε, επίθεση στη βιοπικιλότητα και την ποιότητα του αέρα και ούτω καθεξής, θα χρειαστούμε και περαιτέρω κονδύλια. Και Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές εδώ. Το σύνολο του ελετέ δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα είναι πολύ ψηλότερο από αυτό το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύσκολο θα μπορέσουμε να κρίσουμε τα κράτη-μέλη για αυτό τον προπολογισμό. Και αν τα καταφέρουμε, θα πρέπει πράγματι εντό αυτών των κονδυλίων να υπάρχει και ένα επαναπροσανατολισμό, ο οποίο θα μα επιτρέψει να δούμε ότι ό,τι κάνουμε είναι συντονισμένο για να πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η απάντηση σήμερα σε αυτή την ερώτηση. Συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση, αλλά θα ήθελα να επιστρέψω στις ιδιωτικέ επενδύσεις. Εδώ θα χρειαστεί να υπάρχει και ένα σαφές και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ε, τι ε, είναι βιώσιμη επένδυση. Αυτό όμως ε, δεν είναι μόνο δική σας αρμοδιότητα, την ε, μοιράζεστε με τον ε, Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και με τον Επίτροπο Τζεντιλόνη. Τι θα κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες και θα εγγυηθεί κατάλληλη χρηματοδότηση του Green Deal και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, το θίξατε, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως κλιματική τράπεζα της Ευρώπης και κυρίως όσον αφορά τις επόμενες συζητήσει ε, για επενδύσεις ε, σε ορυκτά καύσιμα. Απάντηση. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπε ο Παύλο Τζεντιλόνι εδώ και ο Βαλτή Ντομπρόσκη ε, σήμερα το πρωί και όλα είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Επομένως ε, υπάρχει πλήρη σύμπνοια επ' αυτού και συμβαδίζουμε. Και αυτό πραγματικά ε, μου δίνει και διάθεση να ξεκινήσω, διότι όπως σας είπα πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και θέλω να αποδείξω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μπορούμε να το κάνουμε. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, ε, Ήδη έχω μιλήσει με τον πρόεδρο τη Τράπεζας Επενδύσεων και ο ίδιο δεσμεύεται ιδιαίτερα για να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η Τράπεζα Επενδύσεων μετά από τι επιτυχίε του σχεδίου Juncker είναι διατεθειμένη να πει επακριβώ τι θέλει να κάνει με τι επενδύσεις που μπορούν να γίνουν και πρέπει να πάνε προ αυτή την κατεύθυνση και για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ε, αποδεσμευτούν από μια ενέργεια που δεν έχει μέλλον. Και εδώ λοιπόν είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτέ τι επενδύσει από του χρόνου, από φέτο, δεν ξέρω πότε ακριβώ, αλλά σύντομα. Thank you for... <coughs> Sorry, for EPP. Ο Γιάννη Κίζα και τώρα έχει το λόγο για το ΕΛΚΑ. Καλησπέρα κύριε Τιμέρμαν, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Ε, ε διάβασα προσεκτικά την επιστολή ε, για την αποστολή σας, ε, τις γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε και ακόμα δεν έχω πιστεί και ακόμα και μετά τα εισαγωγικά σχόλια που μας κάνατε. Ε, είπατε ε, πως θέλετε να επενδυθούν ε, δισεκατομμύρια ευρώ ε, μέσα σε μία δεκαετία και νομίζω πως θα πρέπει να έχετε κάποια επαφή με την πραγματικότητα γιατί δεν πρόκειται να γίνει κάτι αυτό από την πλευρά των κρατών μελών στο πλαίσιο πάντως του Ταμείου της Δίκαιας Μετάβασης. Μετά, επειδή εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Μεταφορών, θεωρείται πως πάντοτε θα πρέπει να υπάρξει ε, περαιτέρω επιβάρυνση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αεροπορία, την αυτιλία και ούτω καθεξής. Ε, εάν θέλετε πράγματι δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα πλέον στον ίδιο βαθμό διαθέσιμα για αυτούς τους τομείς θα ε, ειστρέψουν και πάλι στους ίδιους ε, τομείς με διαφορετικό τρόπο ή θα αναδιατεθούν αλλού. Θα ήθελα δηλαδή να διασφαλιστεί ότι για τους εν λόγω κλάδους η δύναμη της καινοτομία που έχουν, ειδικότερα δηλαδή αναφέρομαι στην αυτιλία και στην αεροπορία, να παραμείνει σε αυτούς και βέβαια αυτό αποτελεί και μια σημαντική προοπτική, μια σημαντική οπτική γωνία ε, για την Επιτροπή Μεταφορών απάντηση. Ε, ναι, εδώ βέβαια το ζήτημα του πόσα κονδύλια θα επενδυθούν στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης ε, είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή μιλάμε ακριβώς για ε, κονδύλια τα οποία θα πρέπει να διατεθούν προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη μετάβαση και σε αυτούς τους κλάδους. Εκείνο που δεν αντιλαμβάνομαι είναι το γιατί θεωρεί κανείς ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με κλάδους όπως αυτός της ναυτιλίας ε, και της αεροπορίας ε, γιατί είναι ήδη επιβαρημένοι. Πώ θα εξηγήσουμε σε έναν καταναλωτή δηλαδή ότι ε, θα πρέπει να καταβάλει φόρου για παράδειγμα για τα καύσιμα όταν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ή θα πρέπει να καταβάλει αντίστοιχου φόρου ε, για το τρένο, αλλά για παράδειγμα για την κυροζήνη ε, δεν είναι απαραίτητο να καταβάλλονται φόροι. Δεν μπορεί να, να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι παράλογο τη σήμερον ημέρα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ειλικρινεί σε ό,τι αφορά τη φορολογική μα πολιτική. Δηλαδή θα ήταν μια διαφορετική πολιτική ε, ωφέλιμη για το σύνολο της κοινωνίας μας. Και ε, νομίζω πως θα ακούσατε στα σχόλια που έκανα εισαγωγικά ότι το ζητούμενο δεν είναι να μην χρησιμοποιούν πλέον τα αυτοκίνητά τους οι πολίτες μας, αλλά να έχουμε αυτοκίνητα ε, τα οποία δεν έχουν αυτές τις εκπομπές όπως τις έχουν σήμερα και νομίζω πως μπορούμε να το επιτύχουμε μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Ή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αφιλία, είδατε πραγματικά ποιες είναι οι εκπομπές, ποια είναι η ρήπανση Εντάξει, κάτι θα πρέπει να γίνει είτε στο επίπεδο του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, είτε αν δεν γίνει εκεί, σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχετε, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μεγέθου πλοίο, για παράδειγμα, στον ε, λιμένα του Αμβούργου, είτε είναι κρουαζιερόπλοιο, είτε κάτι άλλο, ε, βλέπετε πόσο αυξάνεται εκεί η ρήπανση στο λιμένα. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνουμε και κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Δεύτερη ερώτηση. Ναι, πράγματι, το βλέπουμε αυτό και στο Άμστερνταμ και αλλού, σε μεγάλους λιμένους, ε, πράγματι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ε, μετά. Ε, ε, πρόκειται για ένα παζλ, δηλαδή, είπατε ότι θέλετε να, στο, ερώτημα που έθεσε ο Σάλφο Λάγκη, ότι θέλετε να ε, συνεργαστείτε με την Επίτροπο Βεστάγκερ. Ε, ε, θα κάνετε όμως πραγματικά όλες αυτές τις προσπάθειες ταυτόχρονα. Είσαστε τελικά δηλαδή ένας ομαδικός παίκτη αν θέλετε στην Επιτροπή μεταξύ ισοτήμων ή θα είσαστε ο αρμόδιος για όλα αυτά. Και μόνος αρμόδιος. Νομίζω πως έχω καταδείξει ότι είμαι team player πραγματικά και τα όσα αναφέρω σήμερα εδώ πραγματικά <coughs> βασίζονται στην ομιλία της υποψήφιας πρόεδρου της Επιτροπής κ. Φοντρελάιν. Ίσως να το έχετε ξεχάσει. Όχι, εντάξει, δεν το ξεχάσατε, μου λέτε. Ωραία, θετικό είναι αυτό. Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια συνεργάστηκα πολύ στενά με του υπόλοιπου επιτροπού ε, και το είπα και σήμερα το βράδυ εδώ ότι δεν μπορεί κανεί να το επιτύχει μόνο του ω επιτροπό. Θα πρέπει να το κάνουμε από κοινού. Υπό την ηγεσία τη ε, κυρία Ούσουλα Φοντερ Λάιν. Και χρειάζομαι δηλαδή του άλλου επιτρόπου ε, στου διάφορου ε, τομεί, αλλά υπάρχει και αρμοδιότητα εδώ σε μένα σε ό,τι αφορά το να κινούμαστε όλοι προ την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό ισχύει για τι μεταφορέ, ισχύει για την αγροτική πολιτική, ισχύει για την περιβαλλοντική πολιτική. Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των πολιτικών. Και αυτό είναι εδώ το δικό μου καθήκον. Και θα το κάνω από κοινού με του συναδέλφου μου, όπω το έκανα και τα τελευταία πέντε χρόνια με του επιτρόπου. Thank you for GUE. E, Anza Azekamp. Thank you. Κυρία Χάζενκαμ, κύριε Τίμερμαντσε, όταν μιλάμε για το κλίμα, θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να εκπέμπει ρήπου στο σύντομο των δυνατόν. Πολλά άκουσα, αλλά τίποτα συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. Για το γεγονό ότι η κτηνοτροφία παράγει πιο πολλές, ε, πολλά αέρια παρά όλα τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και τα πλοία μαζί. Δεν μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν τίποτα χωρί να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη εντατική κτηνοτροφία ε, στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη κάνει το αντίθετο. Δεν ε, αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, αλλά δίνει επιδοτήσει στην κτηνοτροφία με των αγροτικών επιδοτήσεων. Και αυτό ε, θα σημαίνει μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία και πιο πολλέ εκπομπέ, πιο πολλή αποψήλωση. Η βασική ερώτηση λοιπόν κύριε Τίμερμανς είναι πώς θα μειώσετε την παραγωγή και την κατανάλωση κρέατος. Ε, θα, πώς θα αντιμετωπίσετε τα εκατομμύρια που δίνονται στην ε, βιολογική βιομηχανία και στο, στην πράσινη συμφωνία αυτή. Περιλαμβάνεται και κάτι για την ευημερία των ζώων, γιατί παρά τις ε, ωραίες υποσχέσεις σας, τα τελευταία πέντε χρόνια ουσιαστικά σταματήσατε τη νέα νομοθεσία και τα θύματα ήταν τα ζώα, το κλίμα και είμαι περίεργη να δω τι θα κάνετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Απάντηση. Πείτε μου όμως ποιους κανόνες καθυστέρησα τα τελευταία χρόνια που αποτρέπουν την ευμερία των ζώων. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά να μου πείτε παρακαλώ για την εντατική κτηνοτροφία, ότι είναι τμήμα του προβλήματος, αυτό το ξέρει και ο αγροτικός κλάδος. Το ξέρουν και οι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Το γεγονός ότι η κτηνοτροφία μπορεί να αποτελέσει και τμήμα της λύσης όμως, αυτό θα πρέπει να το σπίσουμε. Και εδώ θεωρώ ότι υπάρχουν πιο πολλές ε, οι δυνατότητες ε, πέρα από την ε, κατάργηση ουσιαστικά ή τη της κτηνοτροφίας. Αυτό υπονοείται νομίζω. Νομίζω ότι καλό είναι να σκεφτούμε και τον κλάδο της ε, δίαιτας ε, και σίγουρα για μένα θα ήταν καλό και καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε τι επιβάρυνση συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον αλλά επίσης νομίζω ότι σωστό είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγροτικό κλάδο για να κάνει τη μετάβαση αυτή σε ό,τι αφορά τι ε, καινοτομίε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι ε, ζωοτροφέ που καταναλώνονται, την εντατική κτηνοτροφία, πώ μπορεί να καταστεί δυνατή αυτή, πώ ε, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός με άλλε μορφέ γεωργία, για να μειωθεί η πίεση στο περιβάλλον. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική. Θεωρώ ότι αλλά και στα τελευταία πέντε χρόνια του συναδέλφου μου, του κ. Χόγκαν, κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και διαπιστώνω ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή για την ευημερία των ζώων από ότι στο παρελθόν. Αυτό οδήγησε και σε αλλαγή στο γεωργικό κλάδο και θέλουν οι κτηνοτροφικοί γεωργοί να είναι τμήμα αυτές της αλλαγή. Δεν θέλω λοιπόν να είμαι απεσιόδοξο. Θέλω να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου αυτό που σήμερα αποτελεί πρόβλημα, εντατική κτηνοτροφία, να εξελιχθεί προς μια κτηνοτροφία η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ε, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και σε ό,τι αφορά και την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκή Υπήρου, την οποία προτιμούμε να την έχουμε στα δικά μας χέρια παρά να την αφήσουμε στα χέρια των διεθνών αγορών. Ερώτηση. Με απογοητεύει η απάντησή σας, ε, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ε, μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά το τμήμα της ε, διατροφής μας που είναι ε, αρνητικό και επιβλαβές για τα ζώα. Να σταματήσουμε να το επιδοτούμε. Γιατί δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να ανησυχούμε για την αποψήλωση του Αμαζονίου και να υποστηρίξουμε την πυρηνική ενέργεια, γιατί θα πετύχουμε πιο εύκολα τους στόχους μας. Αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω γιατί είπατε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε μικρό επίπεδο για το πώ μπορούμε να επηρεάσετε εσεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι Βρυξέλλε επιδοτούν την κατανάλωση κρέατο, αλλά προωθεί και το κρέα αυτό. Το What a Wonderful Beef, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την, το Ισπανικό κρέα. Σκοπεύετε να σταματήσετε τέτοιε επιδοτήσει και προώθηση των προϊόντων αυτών. Όχι. Για να σας πω με πάσα ειλικρινή, όχι. Σκοπεύω να ασκήσω μια πολιτική η οποία θα οδηγήσει σε μια εκτινοτροφία που θα είναι βιώσιμη. Είμαι υπέρ μιας πολιτικής ε, στην οποία θα ληφθεί υπόψη πιο πολύ η ευμερία του ζώου και θα βελτιωθεί η ευμερία του ζώου. Είτε μιλάμε για την εκτενοτροφία, είτε μιλάμε για τη μεταφορά των ζώων, είτε μιλάμε για τη σφαγή των ζώων. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλάβουν οι αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές ως επιτοπλίστων. Και μία παρατήρηση να κάνω. Σταματήστε λοιπόν τις επιδοτήσεις και κάντε το τώρα, λέτε. Φυσικά έχουμε μεγάλο περιθώριο για τη διαμόρφωση των επιδοτήσεών μας και να την προσανατολισμό του σε διαφορετική κατεύθυνση. Αλλά για να σταματήσουμε έτσι απλά τι επιδοτήσει, έχετε καμία ιδέα τι κοινωνικό αντίκτυπο θα είχε αυτό στην ύπεθρο ε, τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σταματήσουμε σε μία νύχτα τι επιδοτήσει. Και αυτό θα πρέπει να, λάβει, να το λάβει υπόψη η ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και εμένα και τους πολιτικούς ευθύνοντες γιατί θα πρέπει ο κόσμο να υποστηρίξει αυτή την αλλαγή. Θα πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται δυστυχώ πάρα πολλοί άνθρωποι στον αγροτικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο Σεπ Ευχαριστώ. Ε. Πίσω σας άλλη μια ερώτηση. Θα ήθελα να επιστρέψω στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το περίγραμμα αυτό που μας προτείνει. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε σενάριο, πέραν του σενάριου 1, ε, δεν θα μας ε, οδηγήσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε ώστε τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν ε, το καθένα να επιτύχει τους δικούς τους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Προβλέπετε κάποια δεσμευτική εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο των στόχων βιώσιμης και πώς θα γίνει αυτό. Και επίση, αναφερθήκατε στη διάσκεψη βιοποικιλότητας ε, στην Κίνα και το στόχο βιώσιμη ανάπτυξης 15 για την βιοποικιλότητα. Τι θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο αν έχουμε κάποιο στόχο δεσμευτικό. Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ε, πώ άλλαξε το σκεπτικό για τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Θυμάμαι πόσο δύσκολο ε, πέρασε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα να έχουμε και τις τρεις εναλλακτικέ εκδοχέ. Τώρα όμως δεν φαίνεται να μιλάει κανεί για τίποτα άλλο πέραν από το σενάριο 1 και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την ερώτησή σας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη δέσμευση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στα κράτη-μέλη που ήγηκε η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσει τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να εφαρμόσετε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και πώς θα τα καταφέρετε, τι σκοπεύετε σε κάθε τομέα. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε να τα καταφέρουμε για τις επόμενες διασκέψεις, ε, είτε για τη διάσκεψη στη Χιλή, ή στην Γλασκόβη ή στην Κίνα τον Οκτώβριο του χρόνου, θα πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι για τα θέματα αυτά. Και ιδίως ε, το πρόβλημα με τη βιοποικιλότητα και εδώ έχω ζητήσει και κάποιε επιστημονικέ ε, συμβουλέ και το είπα και πριν από δύο εβδομάδε στη Νέα Υόρκη. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι το ορόσημό σα. Πώ το ποσοτικοποιούμε. Με τι εκπομπέ είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα, αλλά με τη βιοπικιλότητα είναι πολύ πιο σύνθετο από επιστημονική σκοπιά. Αυτό που θέλω να κάνω λοιπόν είναι να συζητήσουμε με την επιστημονική κοινότητα, να βοηθήσουμε να έχουμε κάποια ερώτημα τα οποία θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ορόσημα, συγγνώμη, τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να βασίσουμε και τις πολιτικές μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε πριν ξεκινήσουμε ε, το οτιδήποτε. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί ένα από του λόγου που δεν επιτυχάνουμε του παρόντε ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη είναι γιατί δεν έχουμε κάποιου απτού στόχου. Ε, όσον αφορά το εσωτερικό θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θεωρείτε ότι η Γενική Διεύθυνση Κλίμα, αν αναλάβει περισσότερα πράγματα για τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ, ε, θα έχουμε ένα πιο λογικό τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ξέρουμε ποιο ακριβώ θα είναι ο στόχο, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου μα. Νομίζω ότι θα ήταν λογικό ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε το διαχωρισμό μεταξύ του τι θα περιλαμβάνει ο πρώτο και τι θα περιλαμβάνει ο δεύτερο πυλώνα. Και αν δείτε και τι διαφορέ ε, στα αριθμητικά στοιχεία, αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Γεωργία να πάμε προ την κατεύθυνση που θέλει να πάει, ο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών από ό,τι έχουμε τώρα. Θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση για την αντιστοιχία μεταξύ των δύο πυλώνων και αν όχι, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ο γεωργικός τομέας να κάνει αυτές τις αλλαγές ε, για να έχουμε και αυξημένες δυνατότητες για το δεύτερο πυλώνα. For the τώρα για τους πράσινους. Κύριε Τιμερμαντς, ε, είπατε ότι θέλετε να υπάρξει περισσότερη έρευνα, αλλά υπάρχουν ήδη τα αποτελέσματα της έρευνας. Ε, για παράδειγμα, η έκθεση του IPCC σε ό,τι αφορά το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Και ποιο είναι το συμπέρασμα εκεί, πολύ ξεκάθαρο, ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση άμεσα, αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Και έχει, αναφέρεται εκεί και ένα συγκεκριμένο προπολογισμό. Και με βάση του υπολογισμού που γίνονται ε, σήμερα, 8 ε, ε, χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να, τα, να επιτύχουμε ε, αυτό που θέλουμε για τον στόχο του 1,5 βαθμού. Οπότε σας ερωτώ, θα κάνετε αυτά που χρειάζεται να κάνετε και σε επίπεδο προπολογισμού για να το επιτύχουμε. γιατί δεν μας δίνετε πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις. Δηλαδή σας ερωτώ πότε ακριβώς θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα ε, ε, τα οποία προτείνεται. Γιατί αυτό θέλουν να μάθουν οι πολιτέ μα, πότε ακριβώ θα αναλυφθεί αυτή η δράση. Και μετά αναφερθήκατε στι διάφορε ε, αντιφατικές πολιτικές, αλληλοσυγκρουόμενες πολιτικέ. Επιχαίρω το γεγονό που το αναφέρατε, γιατί έχετε πολύ δύναμη τώρα. είσαστε μεν την player, ομαδικό επέκτης, αλλά έχετε και ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδου καύσιμα τα οποία δεν είναι βιώσιμα όπως ε, φινικέλο και άλλα, ε, ε, μπορείτε, θα, κάνετε ό,τι μπορείτε και να μειωθεί η χρήση του ώστε να έχουμε πιο βιώσιμα καύσιμα και θα επιβάλλετε φορολογία στην κυροζήνη και στα σχετικά καύσιμα, δηλαδή στην ναυτιλία και θα επιβάλλετε κυρώσει στα κράτη-μέλα τα οποία δεν θα προτείνουν συγκεκριμένα σχέδια δράση ώστε να προβλέψουν τη σταδιακή εγκατάλειψη των ε, ε, καυσίμων. Ναι, νομίζω πω θα χρειαστούμε καλά εργαλεία στη διάθεσή μα και τα σωστά και τους σωστού στόχους αλλά ε, επειδή μου έχετε θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα και προηγουμένω και έχω ζητήσει κάποιε συμβουλέ, να σα πω ότι με βάση του στόχου που έχουμε θέσει, μπορούμε να τα καταφέρουμε στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ειδικότερα αν θέσουμε πιο συγκεκριμένου ενδιάμεσου στόχου. Και για να σα ε, προσθέσω εδώ και έναν ακόμα τρόπο υπολογισμού. Με όλε βέβαια τι αβεβαιότητε οι οποίε υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτού του κινούμενου στόχου μα, αν θέλετε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι πιο περίπλοκο ακριβώς, ακριβώς γιατί θα αποτελέσει εμπόδιο σε ό,τι αφορά την, την επίτευξη αυτών των στόχων, δηλαδή το να έχουμε πιο περίπλοκους ε, τρόπους υπολογισμού τώρα. Ε, νομίζω σε ό,τι αφορά τις αντικρώμενες ε, πολιτικές έχουμε κάνει ε, το σωστό ε, βήμα. Για παράδειγμα, για το φινικέλαιο και τη μη χρήση του και μπορούμε να κάνουμε και περαιτέρω κινήσεις ε, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους προϊόντα έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη δράση για να μην έχουμε περισσότερη αποψήλωση. Ε, όμως για να το επιτύχουμε αυτό θα χρειαστεί να ε, προβούμε και σε ένα διάλογο με τις χώρες προέλευσης αυτών των καυσίμων γιατί εν λόγω χώρες ε, έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, τις δικές τους αξιώσεις σε ό,τι αφορά ε, το δίκαιο εμπόριο στο πλαίσιο της σχέσης τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια από τα κινήματα τα οποία έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, για παράδειγμα στην Ασία, με ενθαρρύνουν. Ε, δηλαδή θα πρέπει πράγματι και εμεί με τον τρόπο μα να ενθαρρύνουμε αυτέ τι χώρε να μην προβαίνουν σε αποψήλωση σε ό,τι αφορά την υποκίνηση τη παραγωγή του. της παραγωγής τους. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία η οποία θα συμβάλλει στην αποφυγή του να συμβάλλουμε στην αποψήλωση. Γιατί σε διαφορετικό τρόπο θα είναι ε, ή μάλλον αυτή η νομοθεσία θα είναι απολύτω απαραίτητη. Τώρα με ρωτάτε πότε ακριβώ θα αναλυφθεί αυτή η δράση και σα λέω το ταχύτερο δυνατό. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολίτε μα ε, ε, θεωρούν πω είναι πολύ έκτακτο το να αναλάβουμε δράση, αλλά από την άλλη πλευρά, αν είμαστε υπερβολικά βιαστικοί, μπορεί να κάνουμε κάτι λάθο και ουσιαστικά να υπονομεύσουμε την προσπάθειά μα. Οπότε αυτό είναι ο για τον οποίο είμαι προσεκτικό. Εάν θέλουμε να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, τότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να κάνουμε όλη την προπαρασκευαστική δουλειά, να κάνουμε όλε τι αξιολογήσει που χρειάζονται, έτσι ώστε να έχουμε πολύ περισσότερη αξιοπιστία και να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι ω προ τον τρόπο με τον οποίο δρούμε. Οπότε, όταν με ρωτάτε πότε θα αναλάβουμε δράση, σα απαντώ μόλι θα είμαστε έτοιμοι. Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό για το διοξείδιο του άνθρακα δεν μου αποδέσατε, αλλά υπάρχει η δηματικη Υπηρεσία Περιβάλλοντο η οποία αναφέρεται ε, σε έναν τόνο διοξιδίου του άνθρακα ε, ω ε, τιμή. Έχει συγκεκριμένη τιμή και αναφέρεται ε, εδώ και συγκεκριμένη τιμή που έχει προταθεί από κάποιους σε ό,τι αφορά ακριβώς τι εκπομπές. Αλλά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά του Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία εκεί. Εσείς λοιπόν θα μπορούσατε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ε, τιμή σε ό,τι αφορά τις, ε, αυτό το flow price στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Τουλάχιστον σε ένα επίπεδο των 40 ευρώ. Και εγώ σας ε, ερώτησα συγκεκριμένα ως προς το πότε ε, τα μέτρα τα οποία θέλετε να προτείνετε θα ε, τεθούν σε ισχύ. Πότε θα έχουμε δηλαδή τις πρώτες μειώσεις ετώνους. Και μετά σε ό,τι αφορά το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, θα υπάρχει ακριβώς δυνατότητα σε ό,τι αφορά την κατάργηση του άνθρακα. Θα προτείνετε κάτι τέτοιο. Ναι, σε ό,τι αφορά την τιμή για την τις εκπομπές. Ε, δεν θέλω να ορίσουμε εμείς κάποιο ε, συγκεκριμένο όριο, θεωρούμε όπως ε, κινείται σωστά και θα συνεχίσει να το κάνει. Τώρα, πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται το τόνο σύστημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτε σε μένα, αλλά το θέτω και εγώ σε εσά. Όταν θα έχει περάσει απαραίτητη νομοθεσία από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και με βάση τη δική μου εμπειρία, ε, όταν κανείς έχει προετοιμάσει σωστά την νομοθεσία και έχει τα απαραίτητα δεδομένα στη διάθεσή του, έχει καλύτερες ε, πιθανότητες να επιτύχει στην προσπάθεια του. Οπότε, εγώ θα βασιστώ στη δική σας ε, υποστήριξη, έτσι ώστε να είμαι φιλόδοξος στα όσα θέλω να επιτύχω, για να ανταποκριθώ στους πολίτες μας για αυτά που ερώτησαν. Ζητώ, συγγνώμη, αλλά ξέχασα το τελευταίο ερώτημα που μου θέσατε. Ναι, αφορά την αεροσιμότητα των κοντιλίων για το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση. Α, ναι. Ε, σίγουρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα όσα κάνουμε δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και μετά, εάν θέλουμε ε, να πείσουμε τους πολίτες μας ότι θα πρέπει τα χρήματα αυτά τα οποία μα δίνουν ω φορολογούμενοι θα πρέπει να διατεθούν για το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, τότε θα πρέπει να του πείσουμε ότι τα όσα κάνουμε είναι σωστά και ότι πράγματι συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Νομίζω λοιπόν ε, πω ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ταμεία τα οποία ε, προβλέπουμε για τέτοιου είδου ε, μετάβαση για τον εξυγχρονισμό τη ευρωπαϊκή οικονομία, δεν υπάρχει πρόβλημα να μειωθούν αυτέ οι αιρεσιμότητε. Για το Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, το σύστημα εμπορίας ρήπων λοιπόν, είναι μια επιτυχία και όλοι οι τομείς έχουν πετύχει του μεμονωμένους στόχους αυτοί που δεν έχουν υπαχθεί στο ETS ε, έχουν προβλήματα. Επίσης, οι εγγύησει ETS ε, μειώνουν τις εκπομπές γιατί ο αριθμός των επιστοποιητικών μειώνεται κάθε χρόνο. Και παρεμπιπτόντως αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν θα το είχαμε με ένα, με φόρο διοξιδίου άνθρακα. Δεν καθορίζει όμως ποιες τεχνολογικές λύσεις θα εφαρμοστούν. Το ETS είναι ένα σύστημα ανοιχτή προσέγγιση και οικονομικό σύστημα για την αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματο και τη ε, αύξηση τη θερμοκρασία. Η οικονομία λοιπόν και η οικολογία θα πρέπει να πάνε χέρι-χέρι προ την κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται όμω περαιτέρω δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί το κλίμα είναι ένα. Συζητήσαμε το θέμα του φόρου για τα σαν φόρο στα σύνορα για, τις, για τη του ανθρακά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο φόρο. Αν συμφωνείτε με την ιδέα αυτή, ποιε χώρε νομίζετε ότι, νομίζετε ότι είναι κατάλληλες ε, η Καναδά, η Καλιφόρνια, ποιες χώρες πιστεύετε ότι είναι... Ε, απάντηση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα τιμωρηθούμε τελικά για τα βήματα που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά τον αγωνισμό, τις ε, χαμηλές τιμέ από άλλε χώρε όπου δεν θα λάβουν μέτρα. Δύο επιλογέ έχουμε. Είτε θα πείσουμε τις χώρε να κάνουν το ίδιο και να τους πούμε ότι κοιτάξτε αν συμμετέχετε και εσείς στο σύστημα εμπορίας ρήπων, λοιπόν, αν φορολογήσετε τον άνθρακα, αν μειώσετε τις εκπομπές, φυσικά θα είσαστε εταίροι μας και δεν θα χρειαστεί διόρθωση σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα στον άνθρακα και αν δεν θέλετε να το κάνετε λυπόμαστε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να διορθώσουμε αυτή την διαφορά για το αποτύπωμα με ένα φόρο. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι συνάδει και με αυτά που ορίζει ο ΠΟΕ. Αλλά νομίζω ότι αυτά πάνε χέρι-χέρι, γιατί η πρότασή μας θα πρέπει να είναι, κοιτάξτε, συμμετέχετε στο ETS, η θα εφαρμόσουμε άλλε τιμέ για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ιδάλω θα χρειαστεί να λάβουμε δημοσιονομικά μέτρα στα σύνορα. Χαίρομαι με την απάντησή σας. Μιλάτε για ανοιχτέ ανοιχτές λύσει λύσεις και προηγουμένως και μιλήσατε για το υδρογόνο και το υδρογόνο όντως είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργεια, αλλά λιγότερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την κινητικότητα. Μια ένα κινητήρε καύση δεν είναι καλό ή κακός, εξαρτάται και με στο κινητήρι αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει λοιπόν στρατηγική για το υδρογόνο. Ρωτώ, θα εργαστείτε για μια στρατηγική για το υδρογόνο, με τι χρονοδιάγραμμα, πότε αναμένετε να σημειώσουμε επιτυχία σε ό,τι αφορά τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Απάντηση. Σίγουρα θα καταρτήσουμε μια στρατηγική υδρογόνου, γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι και ηγετική δύναμη σε αυτό και έχουμε πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου, αν επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή και πιστεύω ότι το υδρογόνο δεν περιέχει απόλυτη ενέργεια όταν αποθηκεύεται. Ιδανικά θα δημιουργούσα μια εταιρική σχέση με την Αφρική, με την Βόρεια Αφρική για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τεράστιες ε, ε, εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας και να μεταφερθεί αυτή, μάλλον να μετραπεί σε υδρογόνο και να μεταφερθεί με υφιστάμενες οδούς. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουν ε, οι αγωγοί αερίου και να γίνουν αγωγοί υδρογόνου, να χρησιμοποιηθούν ε, ε, τα πρατήρια υδρογοποιημένου αερίου. Ας μην ξεχυλιόμαστε. Αν δεν ενσωματώσουμε μια προοπτική για την Βόρεια Αφρική, για την Αφρική γενικότερα για όλα αυτά, θα αποδυναμωθούμε και από την πλευρά αυτή. Το υδρογόνο λοιπόν πιστεύω ότι αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την οικονομία μας. Αν ο κόσμο στην ε, βιομηχανία του Χάλιβα ήδη λέει ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση στην οποία το υδρογόνο θα ήταν η λύση για μια ανταγωνιστική βιομηχανία Χάλιβα, θεωρώ ότι αυτό σημαίνει τεράστιε ευκαιρίε αν αξιοποιηθεί το δυναμικό στο έπακρο. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από τον Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Όπω ε, ε, και άλλοι συνάδελφοι και εγώ δεν είμαι 100% ικανοποιημένο από τι απαντήσει που δώσατε σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική, το σύστημα εμπορία εκπομπών ε, και άλλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μου αρέσει η δέσμευσή σα και το γεγονό ότι είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με τον Επίτροπο του Πρόφηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τη βιομηχανία. Και σε κάθε περίπτωση υποστηρίζω τη γραμμή σα. Ε, ότι δηλαδή σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους ακολουθείτε τα όσα ανέφερε ε, η κυρία Όσαρα Φονταλάνη στην δική τη ομιλία. Δηλαδή θέλουμε το 50% και αν γίνεται το 55% αλλά θα πρέπει να πληρούνται ορισμένε προποθέσει. Αναφερόμαστε πολύ συχνά στην επιστήμη εδώ, στα σχετικά δεδομένα, αλλά η επιστήμη δεν σέβεται και τα σύνορα. Άρα λοιπόν το βασικό σας καθήκον θα είναι να πείσετε τους άλλους εταίρους μας διεθνώς να κάνουν περισσότερα και από δική του πλευρά. Και αναφερθήκαμε πολύ στην Γκρέτα, τον Μπερκάλα. δεν είναι ε, Όμω εκείνη βρίσκεται στην Ευρώπη. Οπότε ε, δεν σα λέω να μεταβείτε στι Ηνωμένε Πολιτείε, σα λέω να επενδύσετε προσωπικό και προσπάθεια έτσι ώστε να πείσετε τι χώρε άλλου. Και σα ρωτώ λοιπόν τι ακριβώ θα κάνετε για να πείσετε. Ε, τι άλλε αυτές χώρε ε, για να αναλάβουν ε, ε, δέσμευση αντίστοιχη με αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Ναι, το είπα ήδη ότι ένα μεγάλο κομμάτι τη εργασία μου θα είναι ακριβώ αυτό, να πείσουμε του διεθνεί μα εταίρου αλλού στον κόσμο. σω κάποιοι να λένε ότι δεν θεωρούν πω θα πρέπει να γίνει κάτι ή θα πρέπει να γίνει με την ταχύτητα που το επιθυμούμε, αλλά ήδη βρίσκονται σε μια φάση μετασχηματισμού. Η βιομηχανία τους ήδη βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού. Οπότε δεν είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξο. Δηλαδή, εκείνο που λείπει συνήθω από την πλευρά εκείνων των χωρών είναι η πολιτική βούληση. Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι το βασικό μα εμπόδιο, τότε η πολιτική ε, ακριβώ επαφή, οι διαπραγματεύσει σε διεθνέ επίπεδο, το να καταδείξουμε ότι λειτουργεί αυτό το μοντέλο ή για παράδειγμα οι ίσοι όροι του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά το εμπόριο μπορούν να μα βοηθήσουν. Δηλαδή, το να του πούμε για παράδειγμα ότι αν δεν υπάρχουν ίση όροι του παιχνιδιού στο εμπόριο μα, ότι δεν θέλουμε τόσο εμπόριο. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να μα βοηθήσουν. Και Επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι όσα συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου είναι σοκαριστικά για όλους μας σε ό,τι αφορά δηλαδή άλλες χώρες. Για παράδειγμα δείτε τις ε, διάφορες πόλεις στην Κίνα, στην πυρωτική Κίνα. Πραγματικά είναι αποκνικτική εκεί η κατάσταση. Επνίγονται από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα για παράδειγμα, ότι από τα 8 εκατομμύρια εδώ ε, στον πλανήτη, το 1 εκατομμύριο θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν το πόσο επίγον είναι να αναλυστεί ε, δράση. Και, ε, συμφωνώ μαζί σας ό,τι αφορά την ανάγκη λοιπόν του να έρθουμε σε αυτές τις επαφέ, αλλά να πω και κάτι ε, το οποίο δεν το λέτε εσεί, αλλά το λένε άλλοι. Επειδή δηλαδή εμεί σε εμά αντιστοιχεί το 9% των εκπομπών, τότε εκείνοι οι άλλοι που έχουν τι περισσότερε εκπομπέ θα πρέπει να αναλάβουν πρώτη δράση. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Αν εμεί δείξουμε ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί, ότι βοηθάει τη βιομηχανία μα, δημιουργεί θέσει εργασία, ε, τότε αυτό θα αποτελέσει και το πιο πιστικό επιχείρημα έτσι ώστε να μα ακολουθήσουν και άλλοι. Και θα κάνουμε μεγάλε προσπάθειε για να το επιτύχουμε, αλλά ε, και θα κάνω ό,τι μπορώ και για τους παίκτες, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το τομέα της βιομηχανίας ε, αλλού, προκειμένου να αναλάβουν δράση από την πλευρά τους. Ε, και εδώ επανέρχομαι στη συμφωνία ε, στην οποία θέλω να την οποία θέλω να κάνουμε, αν θέλετε, ε, ω κοινωνία ολόκληρη σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι πολίτε να θεωρούν ότι αυτό του επιβάλλεται άνωθεν. Αν ε, δηλαδή οι πολίτε θεωρούν ότι και εκείνοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, τότε νομίζω πω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, και το ότι δεν θα μπορέσω ποτέ βέβαια να έτσι απαντήσω 100% στα όσα επιθυμούν οι συντηρητικοί είναι κάτι το οποίο θεωρώ ως ένα κομπλιμέντο. Κύριος Λίζα και πάλι. Ναι είπατε ότι ναι, θα κάνετε προσπάθειες για να υπάρξει συνεργασία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προσπαθείτε να πείσετε και τους πολίτε. αλλά και σε ό,τι αφορά τους διεθνεί διεθνείς είπατε ότι θα είμαστε πιστικοί αν δεν αναφερόμαστε μόνο σε κανόνες και σε νόμους. Οπότε, σε ό,τι αφορά το one in, one out, δεν ήσασταν πολύ ξεκάθαρο. Δεν θα έπρεπε να προβλέψουμε εδώ κανόνες ε, σε ό,τι αφορά ε, το να μην ε, προσπαθούν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν διαφορετικέ τεχνολογίε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι εδώ σε ό,τι αφορά την κατάργηση τεχνολογιών οι οποίε είναι ε, λαβερές για το περιβάλλον. Απάντηση. Ε, ναι, συμφωνώ μαζί σα, αλλά και τα τελευταία πέντε χρόνια όταν εγώ ηγήθηκα αυτή τη ε, ε, task force σε ό,τι αφορά την καλύτερη νομοθεσία, ζήτησα από τι εθνικέ κυβερνήσει, πείτε μα τι ακριβώ θέλετε να καταργηθεί. Το ζήτησα αυτό από όλου, αλλά δυστυχώ ο κατάλογο τον οποίο είχα στο ήταν πολύ μικρό. Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα εκεί ω προτάσει για κατάργηση. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια για καλύτερη νομοθεσία και πιο προσαρμοσμένη στι ανάγκε ε, νομοθεσία και νομίζω με τι αξιολογήσει ε, αντικτύπου και ε, με την αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη νομοθεσία και ήδη την έχουμε. Και νομίζω πω μπορούμε να θεωρήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλού τομείς για να δούμε αν μα εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, η οδηγία για την ενέργεια. Όχι, δεν βρίσκεται στα επίπεδα που θα επιθυμούσαμε και θα πρέπει να την επανεξετάσουμε αυτή την οδηγία. Και θα ήθελα να υπάρξει η δυνατότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να ε, ε, επιβάλλουμε φορολογική και στην κυρωσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτό το κάψιμο θα πρέπει να εξαιρείται από τη ε, φορολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή και ο κλάδος της αεροπορίας θα πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνουμε είτε μέσω φορολόγηση είτε μέσω συμμετοχή στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτηθεί. Είμαι λοιπόν υπέρ τη καλύτερη νομοθεσία και είμαι υπέρ τη κατάρριξη νομοθεσία η οποία είναι παροχημένη ή δεν μα χρησιμεύει πλέον και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και είμαι στο πλευρό σα σε σχέση με αυτή την προσπάθεια. Αλλά βέβαια εκείνοι οι οποίοι αξιώνουν το να υπάρξει κατάρριξη ε, υφιστάμενη νομοθεσία ε, θα πρέπει να είναι και εκείνοι που θα μα προτείνουν συγκεκριμένα ποια, ποια είναι η νόμη που θέλουν να καταργηθούν. Ευχαριστώ. Ωραία. Ήρθε η στιγμή τώρα για τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει περάσει η ώρα, το ξέρω και σίγουρα έχετε καλύτερα πράγματα να κάνετε από το να ακούτε εμένα για άλλα πέντε λεπτά. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα μήνυμα το οποίο ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Και αυτό είναι το εξή. Τα τελευταία 10-15 χρόνια πολύ συχνά έχει γίνει αυτή η συζήτηση τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ορισμένες φορές οδήγησε και σε μια συζήτηση η οποία υποχρέωσε την ε, πλειονότητα των πολιτών ε, σε κάποιο κράτος μέλος να ψηφίσουν ε, υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ λυπηρό. Αλλά είναι και ένα βάρος για μας, γιατί πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες σε τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι ένα τομέα στον οποίο πρέπει να κάνουμε ελάχιστη προσπάθεια για να του πείσουμε είναι ο τομέα ε, τη αλλαγή τη κοινωνία μα ε, και τη ε, μεταμόρφωσή της σε μια βιώσιμη κοινωνία. Αν δείτε τι αναλύσει πάνω από το 90% των Ευρωπαίων επιθυμούν να δράσουμε για να καταπολεμήσουμε την κρίση για το κλίμα. Ε, πάνω από τους 9 στους 10 πολίτες θέλουν να κάνουμε κάτι επ' αυτού. Και αυτό σημαίνει ότι εσείς και εγώ έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε σε τι χρησιμεύουμε πιο συγκεκριμένα να βοηθήσουμε την κοινωνία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη για να μετατραπεί σε μια βιώσιμη κοινωνία που θα έχει τα ενία του κόσμου. Μπορούμε να είμαστε η ηγετική ήπειρος στον κόσμο που θα οδηγήσει τον κόσμο σε ένα λαμπρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ευκαιρία την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ή να χάσουμε τα πάντα τώρα. Διότι το 2050 μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινό ε, μέχρι να το επιτύχουμε, αλλά εάν δεν έχουμε την νομοθεσία σε αυτή τη φυτία, στην επόμενη πενταετία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε τους στόχους του 2030, πολλό δε μάλλον τους στόχους του 2050. Θα είναι αδύνατον. Και αν δεν το πλαισιώσουμε αυτό εντός των πρώτων 100 ημερών της Επιτροπής Φοντερ Λάιεν, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ετοιμάσουμε την ομοθεσία για την επόμενη πενταετία. Στις επόμενες 100 ημέρες λοιπόν, μετά από την 1η Νοεμβρίου, εσείς και εγώ έχουμε συλλογική ευθύνη προκειμένου να ε, το πετύχουμε αν δω τι μας ζητούν τα παιδιά μας, αν δω ορισμένες φορές και το επίπεδο της απελπισίας σε κάποια σκέλη της κοινωνίας μας, αυτή την αίσθηση ότι κανείς δεν είναι υπεύθυνο, έχουμε μπει σε ένα τρένο και δεν ξέρουμε προς τα που οδεύουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ευρωπαϊκές προκλήσεις. Και αν τα καταφέρουμε σωστά στην Ευρώπη, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι στα χέρια σας ε, να τα καταφέρουμε. Και ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω εδώ στα γρήγορα. Ε, βρήκα κάτι στην σε ένα βιβλίο από τον Winston Churchill, το οποίο αξίζει βραβείο Νόμπελ. Έγραψε για την κατάσταση στη δεκαετία του 30 και βρήκε ένα ποίημα για ένα τρένο ε, στη δεκαετία του 1890 το ε, τρένο αυτό είχε ξεκινήσει μια ξέφρενη πορεία γιατί κανείς δεν ήταν ε, στην, στο τιμόνι. Το πείμα έλεγε το εξής. Το, ο βηματισμός είναι θερμός, πλησιάζουν, υπάρχουν σήματα στη νύχτα, μάταια. Ο θάνατος έχει αναλάβει τα ενία αυτού του τρένου και ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει εκεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει εργοδηγός και ότι ακούει τι έχουν να πούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο εργοδηγός γνωρίζει προς τα που οδεύουμε και έχει και ένα χάρτη ο οποίος θα μας επιτρέψει να φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι δικό σας καθήκον και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το επιτύχουμε όλοι μαζί. Και αν το κάνουμε από κοινού, σίγουρα θα μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε ένα μέλλον για την Ευρώπη, για το οποίο τα παιδιά μας θα είναι περήφανα. Σας ευχαριστώ πολύ.